Συνάδελφοι, δεν είμαστε και πολλοί, αλλά ε, θα ε, έρθουν ενισχύσεις, είμαι σίγουρη. Έχουμε πολύ φορτωμένη μερίσια διάταξη, οπότε ας μην καθυστερήσουμε στην έναρξη. Και ε, θα ξεκινήσουμε με μια ακρόαση, σημείο 18 της ημερησίας διάταξης. Ε, αντίκτυπος της, του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου στις κοινωνικές πολιτικές και τις πολιτικές απασχόλησης. Τέσσερις ομιλητές. Θα μου πείτε είναι λίγο παράδοξο να ε, κάνουμε αυτή την ακρόαση τώρα, ενώ στην Ολομέλεια ψηφίσαμε ήδη την έκθεση Λόπε Φοντανιέ για την ετήσια ε, ε, έκθεση περί ανάπτυξης. Γνωρίζουμε ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο δεν ολοκληρώνεται με την ψηφοφορία στην Επιτροπή μας ούτε με το Σύμβολο Κορυφής της Άνοιξης γιατί το δεύτερο τρίμηνο αφιερώνεται στην υπόβολη από πλευράς των κρατών μελών των εθνικών προγραμμάτων ε, μεταρρύθμισης και των προγραμμάτων ε, ανάπτυξης και σύγκλησης ε, που αργότερα θα μετατραπούν σε συστάσεις σαν χώρα. Ε, όλα αυτά εν ώψη του Συμβουλίου του Ιουνίου, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Ιουνίου. Ο πρόεδρος Φαν Ρόμπαϊ, ε, ε, αν το πολιετές πλαίσιο και οι διάφορες εκλογές δεν επηρεάσουν την κατάσταση, θα υποβάλει συγκεκριμένες καινούργιες προτάσεις για την διαδικασία. Τα συμπεράσματα του ε, τη Συνόδου Κορυφή του Δεκεμβρίου σε κάθε περίπτωση έδωσαν μια καινούργια διάσταση στην συζήτηση. Εν μέρη εμεί ε, την εντάξαμε στην έκθεση Λόπε Φοντανιέ, η οποία στην παράγραφο, μάλλον τα συμπεράσματα στην παράγραφο 12 λένε ότι προσθέτουν μάλλον μια απαραίτητη κοινωνική διάσταση στην πραγματική οικονομική ένωση. Χωρίς ε, να ξέρουμε πολύ καλά ακριβώς τι σημαίνει αυτό, αυτή η προσθήκη. Σε αυτό το συνολικό πλαίσιο θελήσαμε, αποφασίσαμε να οργανώσουμε αυτή την ακρόαση έχοντας ε, στο μυαλό μας και μια ε, συζήτηση μεταξύ της ε, Οικονομικής και Επιτροπής και της δικής μας σε ό,τι αφορά τον κοινωνικό αντίκτυπο Ε, της, ε, των ε, προτάσεων της Κομισιόν για την εξυγίανση του προπολογισμού. Πριν δώσω το λόγο στην εισηγήτρια, πριν δώσω το λόγο μάλλον στους ε, φιλοξενούμενους μας, στους καλεσμένους μας, να δώσω το λόγο στην εισηγήτρια. Για να μας θέσει το πλαίσιο στο οποίο θα κινηθεί η ακρόαση. Ο λόγος στην κυρία Βερόνικα Λόπε Φοντανιέ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Είναι πολύ σημαντική αυτή η ακρόαση. Είναι σημαντικό να ακούσουμε τι νομίζουν οι εκπρόσωποι των οργανώσεων των κοινωνικών εταίρων. Οι εκπρόσωποι των οργανώσεων καλύτερα των μικρών επιχειρήσεων. Θα συνεχίσω ισπανικά. Είναι κρίμα που δεν προλάβαμε να διοργανώσουμε αυτήν την ακρόαση πιο νωρί. Ε, ε, είχαμε πολύ χρόνο μπροστά μας για να συντάξουμε την έκθεση, όμως ε, γίνεται αυτή η ακρόαση πριν από το Συμβούλιο Κορυφής του Τη Άνοιξης, το αερι, της Αερινής Συνόδου ε, οπότε μπορεί να μας ακούσουν. Το Συμβούλιο δηλαδή μπορεί να ξέρει ποιες είναι οι θέσεις μας, ποιες είναι οι προτεραιότητές μας ε, και οι δικές μας και των κοινωνικών εταίρων. Στην έκθεση γίνονται, γίνεται λόγος για δύο συγκεκριμένα πράγματα. Την απασχόληση και την ανεργία. Φενός έχουμε μεγάλο αριθμό νέων ανέργων, ανέργων μεγάλης διάρκεια, ε, γυναίκες, ε, ε, ηλικιωμένοι. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε τι πιστεύουν, ποια είναι η άποψη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τι μπορεί να γίνει πραγματικά για να αντιμετωπίσουμε το θέμα της ανεργίας και να αρχίσουμε να δημιουργούμε θέσεις εργασίας. Και δεύτερον, δεύτερο θέμα της έκθεσης ήταν η φτώχεια, όλο και περισσότερη φτώχεια. Δεν είναι δυνατόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση να έχουμε ένα τόσο μεγάλο αριθμό φτωχών. Η στρατηγική Ευρώπη 2020 είχε ως στόχο την μείωση της φτώχειας, την βελτίωση ε, του βιωτικού επίπεδου των ε, πιο των ε, την του πληθυσμού που αντιμετωπίζουν τα περισσότερα προβλήματα, δηλαδή των γυναικών και των παιδιών. Ε, δεν το έχουμε καταφέρει βέβαια αυτό. Οπότε, ποιε συστάσει, ποιε συμβουλέ μπορούμε να δώσουμε στα κράτη-μέλη για να βελτιώσουμε την κατάσταση. Να διευκολύνουμε την ένταξη των ε, οικογενειών που περνούν δύσκολες στιγμές, ε, που επηρεάζονται περισσότερο από την κρίση από ό,τι άλλοι. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Ώρα να ακούσουμε, να ακούσουμε τους καλεσμένους μας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Να προσθέσω και εγώ δύο λόγια. Θεωρώ ότι έχετε έτοιμες τις παρεμβάσεις σας, αλλά να σας υποβάλω και εγώ κάποια ερωτήματα. Υπάρχουν κάποια θέματα που έχουν ξανανοίξει. Ε, σε αυτή την προσπάθεια για μια πραγματική οικονομική και νομισματική ένωση. Υπάρχει το θέμα των συνθήκων ε, του κοινωνικού διαλόγου σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχει ξανανοίξει αυτό το θέμα, έχει ξαναμπεί στο τραπέζι. Ε, έχετε ιδέε για το πώς μπορεί να εξελιχθεί αυτός ο διάλογο. Αν έχετε τις ιδέε, θα θέλαμε να τι ακούσουμε μεγάλο ενδιαφέρον. Λοιπόν, θέλω να δώσω το λόγο στον Ζακ Ντελπλά σας ευχαριστώ που ήρθατε. Είστε οικονομολόγος. Είναι επίκουρος καθηγητής στο, στη σχολή της Τουλούζης και είναι ένας από τους συντάχτες της πρότασής μας α, ε, δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού σταθεροποιητή μέσω ενός μηχανισμού κοινωνικού για την ασφάλιση της ανεργίας ή τα επιδόματα καλύτερα ανεργία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πώς να ανοίξω το μικρόφωνο μου. Merci, Madame la Présidente. Merci, cher Pervenche. Ευχαριστώ αγαπητή Pervenche. Θέλω να σας μιλήσω για την αγορά εργασίας. Πώς μπορούμε να καταπολεμήσουμε την ε, σημαντική ανεργία που έχουμε στην Ευρωζώνη. Και τώρα θα περάσω στα αγγλικά για να απευθυνθώ σε περισσότερους ανθρώπους. Ε, μαζί με διάφορους άλλους συντάκτες έχω ετοιμάσει αυτό το έγγραφο και δεν είμαστε οι πρώτοι που προτείνουμε ένα μηχανισμό ε, για την καταπολέμηση της ανεργίας στην Ευρωζώνη. Χρειαζόμαστε κάποιες μεταφορές ε, πιστώσεων στην Ευρωζώνη για να αντιμετωπίσουμε τα, τις πιέσεις, τα σοκ. Ε, η Πορτογαλία, η Ελλάδα ε, δεν μπορούν να απορροφήσουν από μόνες τους αυτά τα ασύμετρα σοκ, τις ασύμετρες πιέσεις. Υπάρχει πραγματικά ανάγκη για μεταφορές από τις ευημερούσες ζώνες προς τις μειονεκτούσες ζώνες της Ευρωζώνης. Το θέμα είναι πώς θα γίνει αυτή η ιστορία, ούτω ώστε να μην υπάρξει διάσωση. Και για να το πω έτσι σχηματικά. Εσείς... Όσοι θέλουν, όσες χώρες Ευρωζώνης θέλουν να έχουν ένα τέτοιο μηχανισμό ασφάλισης ανεργίας, γιατί έχουν τεράστιες α, δυσκολίες. Είναι κυρίως οι ζώνες της περιφέρειας, του Νότου, ενώ οι βόρειες χώρες δεν θέλουν, είναι πρόθυμες. Πώς θα πιέσουμε όλους να συμμετάσχουν. Η καινοτομία δεν είναι να έχουμε ένα επίδομα ενεργείας σε όλη την Ευρωζώνη, αλλά να έχουμε κίνητρα ούτω ώστε αυτό το μηχανισμό να το δεχτούν όλοι. Η πρότασή μας ε, βασίζεται σε τρεις πυλώνες. Και οι τρεις χρειάζονται. Ο πρώτος, που είναι απλός, δεν είναι καθόλου καινοτόμος, είναι να βρούμε τους πόρους που προκύπτονται από τις, προκύπτουν συγγνώμη, τις εθνικές α, κοινωνικές πολιτικές. Και με μία κλίδα, ας πούμε, κατανομής, ε, συμμετοχής, ε, κάθε χώρα θα συμμετέχει με το 1% του ΑΕΠ της, σαν ένα κοινό μηχανισμό ασφάλισης της ανεργίας, μιλάμε για όλες τις χώρες της Ευρωζώνης. Αυτός ο μηχανισμός συνδέεται με το ευρώ, έτσι. Αφορά λοιπόν τις χώρες της Ευρωζώνης αποκλειστικά. Και κάτι πολύ σημαντικό μπορούμε να προσθέσουμε την συνιστόσα της κατάρτισης για τους ε, εργαζόμενους. Δηλαδή, η κάθε μία από τις 17 χώρες Ευρωζώνης θα αφιερώσει το ένα, ας πούμε, ή ένα και κάτι, τα 100 του ε, ΑΕΠ της για την ανεργία, για αυτό το μηχανισμό ασφάλισης ανεργίας και αυτός ο μηχανισμός θα εποπτεύεται από την, είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο δεύτερος πυλώνας είναι πιο καινοτόμος. Θέλουμε να δημιουργήσουμε ε, μία Ευρωπαϊκή Σύμβαση Εργασίας. Την ίδια για όλους τους Ευρωπαίους. Την ίδια για όλες τις χώρες. Για όλους τους τομείς, για όλους τους κλάδους. Αλλά θα είναι προαιρετικός αυτός ο μηχανισμός και θα επανέλθω σε αυτό. Σε κάθε χώρα θα έχουμε ε, αυτή τη σύμβαση του νη αυτή τη στιγμή στη χώρα μου έχουμε 17 είδη συμβάσει εργασία. Θα έχουμε 18η δηλαδή. Στην Ιταλία, στην Ισπανία έχουμε 33. Οπότε θα γίνει 34η σύμβαση. Συν όλες οι άλλε. Αυτή την ε, σύμβαση θα την ε, σχεδιάσουμε εδώ στις ε, Βρυξέλλες με τους συνήθεις υπόπτους. Μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ξέρετε τα θεσμικά αυτά μαγειρέματα πολύ καλύτερα από μένα. Και θα χρησιμοποιήσουμε την εμπειρία όλων. Και κανείς εδώ και ειδικά στον Νότο που το χρειάζεται περισσότερο, ε, δεν ξέρει πώς να μεταρρυθμίσει την αγορά εργασίας, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μόνο οι Βόρειοι, Σκανδιναβοί, ε, Δανείοι και Σουηδοί ξέρουν. Ενώ εμείς εδώ οι Νότιοι δεν ξέρουμε. Επομένως πρέπει να είμαστε Ταπεινή, με ταπεινοφροσύνη να προσεγγίζουμε το θέμα. Οποτεδήποτε γίνεται μια απόπειρα στην Ισπανία, α πούμε, είτε στην Ιταλία τέτοιου τύπου, ε, επειδή δεν υπάρχει εμπιστοσύνη, η μεταρρύθμιση αποτυγχάνει. Ανάμεσα στους ε, εργαζομένους και στου εργοδότες υπάρχει δυσπιστία. Με τη διαβούλευση, με τις ε, ευρωπαϊκές οργανώσεις εργοδοτών και εργαζομένων μπορούμε να προσπαθήσουμε να σχεδιάσουμε το, την καλύτερη δυνατή σύμβαση που θα αφορά όλους τους κλάδους, όλες τις χώρες και θεωρούμε ότι και οι βόρειες χώρες θα πιέσουν για ευελιξία και οι νότιες χώρες θα πιέσουν για ασφάλεια. Επομένως έχουμε ένα σχήμα ευέλιξη ασφάλειας εν είδη συμβιβασμού που μοιάζει τόσο πολύ μετά όσα ξέρουμε εδώ στην Ευρώπη. Ο τρίτος πυλώνας που είναι ίσως ο πιο καινοτόμος στην πρότασή μας είναι ότι αυτή η σύμβαση θα είναι προαιρετική. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, όπως είπα, να έχουμε μια ε, σωστά λειτουργούσα αγορά εργασίας ε, σε εθνικό επίπεδο. Ε, έχουμε τις επιχειρήσεις εναντίον των σωματείων, ε, των συνδικάτων και αντίστροφα. Η ιδέα είναι να αποκεντρώσουμε την απόφαση για την ευελιξία στο άτομο, δηλαδή να τη μετακυλήσουμε στο άτομο. Αυτή προαιρετικά όμως. Δηλαδή, ουσιαστικά τι λέω. Αν η Περβάνς Μπερές με προσλάβει στη μικρή της εταιρεία στη Γαλλία. Θα συζητήσουμε το είδος της δουλειάς, της σύμβασης ε, που θα κάνω, ε, της σύμβασης που θα συνάψω κτλ η εταιρεία υποχρεούται να μου παρουσιάσει δύο είδη συμβάσεων τη στιγμή τη υπογραφής. Το πρω... Η πρώτη σύμβαση θα είναι η κλασική εθνική σύμβαση με βάση την ισχύουσα εθνική νομοθεσία, κοινωνική ασφάλιση κτλ. χωρίς καμία αλλαγή, ό,τι ξέρουμε μέχρι στιγμής. Η δεύτερη σύμβαση που θα είναι και αυτή επιτάπητος μπροστά μου θα είναι για την ίδια δουλειά ε, μια Ευρωπαϊκή Σύμβαση εργασία. Ε, με αυτό το πλαίσιο ευέλικτη ασφάλεια, όπως περιέγραψα πριν. Και η ασφάλεια που προσαρτάται είναι, ε, πρώτον θα έχουμε την εθνική ε, πολιτική ασφάλισης, ασφαλίσεων και έξτρα την ευρωπαϊκή πολιτική για τα επιδόματα ανεργίας κτλ. Αν επιλέξω από μόνος μου περισσότερη ευελιξία σε αυτή τη σύμβαση, τότε θα πάρω περισσότερη ασφάλεια σε περίπτωση που με απολύσουν. Η απόφαση για την ευελιξία δεν εξαρτάται από την εταιρεία, αλλά από μένα. Από μένα που υπογράφω τη σύμβαση. Δεν υπάρχει καμία υποχρέωση όμως να την υπογράψω. Οι ιδιότητε τώρα αυτής της σύμβασης είναι σημαντικές. Αυτές οι ασφάλειες είναι πολύ σημαντικές είναι να αποπολιτικοποιήσει όλη τη συζήτηση για τη μεταρρύθμιση της ε, αγοράς εργασίας. αν πάρετε την ε, Ισπανία που είναι η πιο σημαντική ορολογιακή βόμβα αυτή τη στιγμή στην ε, Ευρώπη και η Ελλάδα, ε, τμήμα της ανεργίας είναι διαρθρωτικό, τμήμα είναι κυκλικό. Δεν θέλω να μπω σε πολλές λεπτομέρειες, αλλά υπάρχουν προτάσεις που ασχολούνται αποκλειστικά με την κυκλική ανεργία. Η ευρωπαϊκή ασφάλιση αυτή, αυτό το σχήμα για το οποίο σας ε, μίλησα, θα εξασφαλίσει κάθε εργαζόμενο εναντίον απέναντι στην ε, κυκλική ανεργία. Η ιδέα είναι να παρακάμψει τις τοπικές δυσκολίες και θα του δώσει χρήματα, μάλλον και θα δοθούν χρήματα μόνο αν γίνει ε, δεκτή η μεταρρύθμιση. Στις Βρυξέλλες τώρα γίνονται πολλές συζητήσεις για διάφορες πολιτικές που προωθούν τις εργασίες που βασίζονται σε συμβάσεις. Σύμβαση για παροχή υπηρεσιών. Ε, η Σύνος Κορυφής του Δεκεμβρίου εμεί πρότεινε κάποια πράγματα για αυτές τις συμβάσεις, αυτό προτείνουμε εμείς και πιστεύω ότι η δική μας πρόταση είναι ένα μακροεργαλείο για να αντισταθμίσει την ύφεση και είναι ανώτερο από τις μακροπολιτικές που μου δίνουν απλώς λεφτά επειδή βρίσκομαι σε ύφεση. Εδώ θα έχουμε μια μετακίνηση χρημάτων και δεύτερον θα έχουμε εκτός από αυτό και μεταρρυθμίσεις επιπλέον. Σας ευχαριστώ για αυτές τις σκέψεις είναι πραγματικά τροφή προσκέψη. Ε, ε, Δίνω το λόγο στην Γκουνίλα ε, Άνγκρεν, πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Για 7 λεπτά. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Αγαπητές και αγαπητοί κυρίες και κύριοι. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση που μας απευθύνατε. Ως ε, πρόεδρος της ΟΕΑΜΠΕ που εκπροσωπούμε τους ε, εργοδότες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και εγώ η ίδια επιχειρηματίας ε, που απασχολώ τρεις εργαζόμενους στη Σουηδία θέλω να υπογραμμίσω ότι η πραγματική οικονομία πραγματικά επλήγει από την οικονομική και χρηματοοικονομική κρίση. Το δικό μας ε, βαρόμετρο μικρομεσαίων επιχειρήσεων επιβεβαιώνει ότι οι πολιτικοί λιτότητες και τα μέτρα εξυγίανσης επηρέασαν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης περισσότερο από άλλες επιχειρήσεις. Το, ε, η εμπιστοσύνη των επιχειρηματιών στο, για, στο μέλλον έχει πέσει. Παρόλο το δύσκολο περιβάλλον, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ήταν και εξακολουθούν να παραμένουν βασική πηγή θέσεων εργασία. Στην Ευρώπη αντιπροσωπεύουν το 98% των, ε, του των επιχειρήσεων και παρέχουν τα 2 τρίτα των θέσεων εργασία. Ε, παρόλη την κρίση εξακολουθούν να δημιουργούν θέσει εργασία, αλλά όχι σε όλου του τομεί και γενικότερα με χαμηλότερου ρυθμού από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ε, οι μικρές και μετακινούμενες επιχειρήσεις, ε, ε, δεν είναι πρόθυμες να απολύουν εργαζόμενους για διάφορους λόγους. Πρώτον, γιατί είναι δύσκολο να βρουν ξανά ε, εργατικό δυναμικό ε, με τα κατάλληλα προσόντα και δεύτερον είναι δύσκολο αυτό να γίνει χωρίς να επηρεαστούν η λειτουργία τους. Ταυτόχρονα οι μικρές επιχειρήσεις ε, δεν είναι διατεθειμένες να κάνουν καινούς επενδύσεις, να κάνουν καινούς προσλήψεις μέχρι ότου σταθεροποιηθεί η οικονομική κατάσταση. Αυτά τα πορίσματα επιβεβαιώνουν αυτό που δείχνουν όλες οι στατιστικές, ότι η ανεργία αυξάνεται σταθερά από τα μέσα του 2011 και έχει φτάσει τα ιστορικό, το ιστορικό μάξιμου του 10% το 2012, με μεγάλη αύξηση στην μακροχρόνια ανεργία. Ταυτόχρονα η Ευρώπη μετρά 2 εκατομμύρια ανέργους, κάτι που ε, δείχνει ένα μόνιμο πρόβλημα, ε, μια αντιστοιχία των δεξιοτήτων με τις θέσεις ε, θα πρέπει να παραδεχτούμε ότι το 2012 ήταν ένα, ένα πολύ καλό έτος. Όμως ε, η τάση δείχνει μια ε, αύξηση του χάσματος μεταξύ χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή μεταξύ Βορρά και Νότου κυρίως και αυτό είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό. Μάλιστα χώρες οι οποίες έχουν ήδη εφαρμόσει μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας πριν την κρίση και έχουν πιο ισχυρά ε, συστήματα κοινωνική ασφάλισης θα πάνε καλύτερα. Ε, απ' την άλλη μεριά υπάρχουν χώρε οι οποίε πιο πρόσφατα έχουν κάνει μεταρρυθμίσεις και αυτέ αρχίζουν να βλέπουν μια βελτίωση σε ό,τι αφορά την ανταγωνιστικότητά του, την ανάπτυξη, όπως για παράδειγμα η Ιρλανδία και η Ισπανία. Όμως ε, οι μεταρρυθμίσεις δεν μεταφράζονται αυτόματα σε περισσότερες θέσεις εργασίας, γιατί γνωρίζουμε ότι η απασχόληση προσαρμόζεται πιο αργά δεδομένων των ιδιαιτεροτήτων της αγοράς εργασίας. Η βασική δυσκολία είναι να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη και να αρχίσουμε να αυξάνουμε τις θέσεις εργασίας. Ε, τώρα, το πώς σε σχέση με τη σύνδεση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου με, με τον κοινωνικό πυλώνα δεν είναι τόσο εύκολο. Κανείς θα μπορούσε να πει ότι τα μέτρα λιτότητες και οι περικοπές ε, χειροτέρευσαν το, την, τους δικες και την κοινωνική κατάσταση. Είναι σωστό αυτό για τον κρατικό τομέα, αλλά αυτό ήταν απαραίτητο. Ε, το να επισκυριζόμαστε ότι η κατάσταση ήταν καλύτερη αν δεν είχαμε ε, λάβει μέτρα εξυγίανσης ε, είναι τρελό. Η αύξηση των ε, χρεών θα οδηγούσε σε αύξηση των επιτοκίων και μείωση των επενδύσεων. Η, οικονομική, η χρηματοοικονομική κρίση έγινε οικονομική και κοινωνική κρίση. Όμως το κόστος της αδράνειας θα ήταν ακόμα υψηλότερο. Το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο που έχει ως στόχο την, τον καλύτερο συντονισμό των μακροοικονομικών, κοινωνικών, πολιτικών και πολιτικών απασχόλησης είναι πιο σημαντικό τώρα πια, δεδομένου ότι η κρίση είναι πολυδιάστατη πλέον η ετήσια έκθεση ανάπτυξης ε, αναφέρει ότι πρέπει να αποφύγουμε μακροοικονομικές ανισορροπίες και οι ανακράτος συστάσεις είναι το κατάλληλο, ο κατάλληλος τρόπος για να προωθήσουμε την ανάπτυξη και την απασχόληση στην Ευρώπη. Η δημοσιονομική εξυγένση και η μείωση των κρατικών χρεών είναι απολύτως απαραίτητες για την αύξηση ανταγωνιστικότητας αλλά όχι αρκετά μέτρα. Θα πρέπει να υποστηρίζονται από διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις κυρίως στην αγορά εργασίας. Γι' αυτό το λόγο η Ένωσή μας καλωσορίζει θερμά την συνέχεια που ε, ε τον, τη συνέχεια των προτεραιοτήτων για το 2013 με συνέχιση των μέτρων δημοσιονομικής εξυγίανσης ε, ανάκτηση ε, της δυνατότητας δανεισμού ιδιαίτερα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις από τις τράπεζες προώθηση της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας για σήμερα και για αύριο μέσω βελτίωσης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης της έρευνας και ε, της ανάπτυξης καθώς ε, ε, της καινοτομίας καθώς επίσης και των επενδύσεων σε αυτές. Εξυγχρονισμός της κρατικής διοίκησης Όλε αυτέ οι προτεραιότητε είναι πολύ καλά ισορροπημένε, λαμβάνουν υπόψη την ανάγκη δημοσιονομική εξυγίανση, αλλά ταυτόχρονα αναγνωρίζουν την ανάγκη να προωθηθεί η ανάπτυξη μέσω μακροπρόθεσμων επενδύσεων. Εν ώψη του 2012 ε, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προχώρησε σε ένα ε, δημοσιονομικό σύμφωνο ε, για να ενισχύσει τα μέτρα εξυγίανσης. Όμως αλλά ακόμα δεν έχει εφαρμοστεί η ανάπτυξη καινούριε θέσει εργασία θα πρέπει να, να επιτευχθούν από τον ιδιωτικό τομέα. Η ανάκτηση τη εμπιστοσύνη, ε, για παράδειγμα, μπορεί να γίνει μέσω τη ανασύσταση του ε, τραπεζικού τομέα. Χρειάζονται επίση μεταρρυθμίσει στην αγορά εργασία για τι καινούριε επιχειρήσει. Ε, χρειάζονται μέτρα για να προωθηθεί η, <coughs> η αντιστροφή του κλίματος είναι πολύ σημαντικό να είμαστε, ε, ή μάλλον οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι παρούσε σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και γι' αυτό το λόγο είναι πολύ σημαντικές. Οι, μακροπρόθεσμε επένδυσει μακροπρόθεσμες επενδύσεις για την ανάπτυξη θα πρέπει να συνοδεύονται από προτάσεις, από προσπάθειες για την ενίσχυση της ε, ε, εξυγίανσης. Υποστηρίζουμε θερμά την διάκριση ανάμεσα στην δημοσιονομική εξυγίανση και τις ε, προσπάθειες που θα λαμβάνουν χώρα, ε, ε, περισσότερο υπόψη της ιδιαιτερότητας κάθε κράτους μέλους. Στο πακέτο για την απασχόληση που παρουσιάζει το 2012 είναι καλό και θα πρέπει να γίνουν προσπάθειες για την αναθεώρηση τη μεταρρύθμιση των αγορών εργασίας. Όλες αυτές περιλαμβάνονται στα πλαίσια μεταρρυθμίσεων τα οποία θα ακολουθηθούν από συστάσεις σε εθνικό επίπεδο. Ε, και θα ακολουθηθούν από μια ε, παρακολούθηση της εφαρμογής τους. Το ευρωπαϊκό εξάμεινο θα πρέπει να συνδυαστεί με μια καλύτερη μακροοικονομική και κοινωνική διακυβέρνηση, με μεγαλύτερη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων σε όλα τα επίπεδα συμπεριλαμβανομένου και του ευρωπαϊκού. Επιπλέον, ο προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι μοχλό για την προώθηση μακροπρόθεσμων επενδύσεων και την καταπολέμηση τη ανεργία. Στην σημερινή κατάσταση, η ανάπτυξη θα πρέπει να προέλθει από τον ιδιωτικό τομέα, όπου οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι ατμομηχανή. Οι ευρωπαϊκέ μικρομεσαίες επιχειρήσεις βασίζονται κυρίως στη ζήτηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό το λόγο ε, μπορούμε να ε, πετύχουμε μόνο αν αλλάξουμε το κλίμα και ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη των οικοκυριών και των ιδιωτικών επιχειρήσεων. Ευχαριστώ πολύ. Γιώργεν Νούνιος major Γενικός ε, Γραμματέας του Καρίτας Ευρώπα. President, members of the Euro μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίε και κύριοι, σα ευχαριστώ πάρα πολύ που κάλεσατε την κάρτα σε Europa για να παρουσιάσουμε τι θέσει μα σε ό,τι αφορά τον αντικτύπο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, σε ό,τι αφορά τι ε, πολιτικέ, τι κοινωνικέ και τι ε, πολιτικέ ε, απασχόληση. 49 οργανώσει 46 ευρωπαϊκών χωρών εκπροσωπούμε, σε παγκόσμιο επίπεδο 160 χώρε εκπροσωπούμε δίνοντας βοήθεια σε θύματα της φτώχειας σε όλη την Ευρώπη. Και 23 ε, ε, οργανώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, δραστηριοποιούμαστε. Το Μάρτιο και τον Ιούνιο του 2010 όλα τα κρατημέλη προσυπέγραψαν τους στόχους του 2020. Πάντα τις λαμβάνουμε υπόψη αυτές τις καταφυντήριες γραμμές και κοιτάμε και τις αιτήσεις εκθέσεις, ανάπτυξης και τις συγκρίνουμε με την καθημερινή ζωή. Και κάνουμε μια σχετική έκθεση την οποία έχετε στους φακέλους σας που σας διανεμήθηκαν και που μπορείτε να βρείτε έξω από την είσοδο. Κάνουμε λοιπόν κάποια σύγκριση σε ό,τι αφορά τους τομείς όπου υπάρχει έντονη εμπλοκή του ανθρώπινου στοιχείου στην ε, παιδεία, στην ε, απασχόληση και κυρίως στη μείωση της ένδυας και σε ό,τι αφορά τους ε, στόχους αυτούς, τους τομείς αυτούς, μία λέξη θέλω να πω και να τονίσω, άμεσα χρειαζόμαστε βοήθεια. Στην Caritas Europa ε, αντιμετωπίζουμε καταστροφές ε, και αυτή η καταστροφή έχει να κάνει, είναι ανθρωπογενής. Ε. Μετά από το κύμα μέτρων λιτότητας, ο αντίκτυπος που υπέστη ο κοινωνικό ιστός της Ευρώπης έχει πολλαπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια και θα πρέπει άμεσα να δράσουμε για να σταματήσουμε την τάση αυτή. Ξέρουμε, ξέρετε τι εννοώ η ανεργία των νέων στην Ελλάδα, στην Ισπανία είναι 60% και στις πιο πολλές ευρωπαϊκές χώρες αυξάνεται δραματικά η ένδια και η ενεργεία. Η Κάρτας ε, ζητά την βοήθεια, μάλλον δέχεται αιτήματα βοήθειας από επιχειρήσεις, από ε, μετανάστες, από μικρά παιδιά, από οικογένειες οι οποίοι ε, σε πολλές περιπτώσεις δεν δικαιούνται καν επιδόματα επειδή έχουν επιβληθεί μέτρα λιτότητας και άρα ε, κάνοντας συγκρίσεις με προηγούμενα χρόνια, βλέπουμε πώς ε, εξελίσσονται τα μέτρα ένδυας και πώς περικόπτονται τα σχετικά επιδόματα. Το ευρωπαϊκό εξάμεινο είναι καθεαυτό ένα καλό εργαλείο. Δεν έχει όμως νόημα όσο παραμένει σε επίπεδο μη συγκεκριμένο, μη σαφές σε ό,τι αφορά τη μετάφραση του σε μέτρα αντιμετώπισης της ένδυσης. Τα μέτρα για την ε, λιτότητα σχετίζονται με την Ένδια. Μάλλον φαίνεται ότι τα, ε, η ειδήσια έκθεση αναγνωρίζει ότι η λιτότητα προκαλεί αύξηση της ένδυας, αλλά δεν το αναγνωρίζει αυτό και δεν ε, χρησιμοποιεί το πλήρες δυναμικό του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου οι σχετικές ε, συστάσεις για τα προγράμματα για την μεταρρύθμιση των κρατών μελών, απευθύνονται σε αυτά τα θέματα μόνο περιθωριακά. Θα πρέπει να δούμε τι γίνεται στην, ε, με την κρίση. Μάλλον την προηγούμενη εβδομάδα στο Δουβλίνο παρουσιάστηκε τι γίνεται με πέντε χώρες της, ε, της Ευρώπης. Και επιδεικνύονται ε, τα, οι επιπτώσεις της ε, λιτότητας στους πιο ευάλωτους πληθυσμούς. Και στην έρευνα αυτή καταδεικνύεται ότι 7 χρόνια πριν από την ολοκλήρωση του, των στόχων της 2020, ε, απέχουμε παρασάγκας από τους στόχους αυτούς. Θα πρέπει να προσέξουμε, γιατί αυτοί οι άνθρωποι απομακρύνονται από την αγορά εργασία και από την κανονική κοινωνική ζωή. Είναι εύκολο πλέον σήμερα κανείς να μπει στον κύκλο αυτό της ένδυας και της ανεργίας, αλλά είναι πολύ δύσκολο να βγει από αυτόν τον κύκλο, από αυτό το φαύλο κύκλο. Και υπάρχουν καινούργια δόγματα στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο για την Κυρία, τα οποία δεν έχουν να κάνουν τίποτα με το 2020. όπω ε, όπως για παράδειγμα ότι δεν θα πρέπει καμία τράπεζα να αποτύχει, δεν θα πρέπει, θα πρέπει να υπάρχει λιτότητα. Τα δόγματα αυτά μας οδηγούν σε αυτό που στην κάρτα ε, βλέπουμε καθημερινά, τη σκληρότητα. Για να σωθεί μια τράπεζα ξεσπιτώνεται ε, μια οικογένεια με μικρά παιδιά που ενδεχομένως να οδηγηθεί στην αυτοκτονία γιατί δεν έχει σπίτι μετά να ζήσει. Αυτό πώς βοηθάει την Ευρώπη να εξελίξει από την κρίση. Αυτό ζητάμε να μας πείτε και να κάνετε ε, από την Κάριτας, να υπάρχει συνεκτικότητα μεταξύ της θεωρίας και της πολιτικής σε ό,τι αφορά τους στόχους του 2020. Η έκθεση της ανάπτυξης θα πρέπει να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ε, εκάστοτε προκλήσεις και να βρίσκει και τρόπους αντιμετώπισης του. Τα προγράμματα τα εθνικά για τη μεταρρύθμιση των κρατών μελών θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Αυτά θα πρέπει να είναι τα νέα δόγματα για να μην χαθεί μια ολόκληρη γενιά. Γιατί καμία προσπάθεια δεν είναι υπερβολικά μεγάλη όταν πρόκειται για τη δημιουργία θέσεων εργασία για του νέου και κανένας, ε, καμία προσπάθεια δεν είναι υπερβολικά μεγάλη όταν πρόκειται για το σπάσιμο του παύλου κύκλου αυτού που καταλήγει στην απόλυτη ένδυα παιδιών. Εμείς στην Κάρτας Ζητούμε μόνο από τα κράτη-μέλη και από τους ε, ηθήνοντες να κάνουν αυτά που αποφάσισαν και υπέγραψαν το 2010 να ε, φροντίσουν προκειμένου οι στόχοι του 2020 να καταλήξουν σε σταθεροποίηση της Ευρώπης και όχι ε, αντίθετα ανάποδα. Θα πρέπει να υπάρχει και επιρροή των Εθνικών Κοινοβουλίων από πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε έτοιμοι να δράσετε άμεσα. Ευχαριστώ. Ο Κλοντ Μανουέλ Τριόμφα, που είναι διευθυντή τη οργάνωση Travail et Emploi Europe Société, Association Travail et Emploi Europe Société, δηλαδή, που έχει το ακρονίμιο Άστρες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η οργάνωσή μας ε, περιέχει ε, συνδικάτα, επιχειρήσεις, ε, εμπειρογνώμονες, ακαδημαϊκούς και επί 10 χρόνια ε, μαζί με τους εταίρους της στην Ευρώπη προωθεί διάφορα προγράμματα για την ανδιάφραση των επιχειρήσεων, για τη μεταρρύθμιση των δικαιωμάτων στον χώρο της εργασίας, τον κοινωνικό διάλογο και μέσα σε αυτό το πλαίσιο, μέσα σε 7 λεφτά, θα προσπαθήσω να πω δύο-τρία πράγματα για την επίπτωση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου στις κοινωνικές πολιτικές. Πρώτη παρατήρηση. Αυτή η προσπάθεια είναι εξόχως διαφορετική από τις προηγούμενες προσπάθειες. Όταν ρωτάω τους εταίρους μου στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, η απάντηση η πιο εύκολη που μου δίνουν είναι όχι. Στα χαρτιά ε, συγκεντρώσαμε τις διαδικασίες, τις ομαδοποίησαμε, αλλά τελικά σε επίπεδο περιεχομένου, σε επίπεδο συντονισμού και μεταξύ των κρατών και μεταξύ των πολιτικών έχουμε σημειώσει μεγάλα βήματα. Προς το παρόν και για να μην σκοτώσω τα πράγματα εν το γεννάστε και να μην είμαι από την αρχή απεσιόδοξο θα πω ότι τίποτα τέτοιο δεν ε, διαφαίνεται. Δεν υπάρχει κάτι τουλάχιστον απτά. Έτσι η όλη προσπάθεια, οι σοσιαλιστές και το ΕΛΚ είναι σε μεγάλες διαπραγματεύσεις. Το καταλαβαίνω, καταλαβαίνω ότι εσείς έχετε τα δικά σας ε, πηγαδάκια, αλλά έχουμε μια ακρόαση εδώ πέρα ένα εξελίξη, που είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Εντάξει, ό,τι θέλετε κάνετε, αλλά σας παρακαλώ. Ο μιλητής ξανά που τον διάκοψε η Πρόεδρος. Λοιπόν, για το περιεχόμενο είναι καλό να κάνουμε μια εγκάρσια ανάλυση των συστάσεων της Κομισιόν προς τα διάφορα κράτη-μέλη σε ό,τι αφορά την, τις πολιτικές απασχόλησης και τις κοινωνικές πολιτικές, όπου υπάρχει ένα έντονο στοιχείο και κυρίως θα σταθώ στις πολιτικές απασχόλησης, τις ξέρω καλύτερα από τις κοινωνικές πολιτικές εν γέννη. Και θα πω ότι όλες βασίζονται σε μία υπόθεση ότι η ανταγωνιστικότητα περνάει μέσα από τις διαφορετικές μεταρρυθμίσεις της αγοράς εργασίας. Όμως, να, να κάνω δύο παρατηρήσεις που συζητάμε στο δίκτυό μας. Πού είναι οι αποδείξεις αυτού του δόγματος. Εδώ και δέκα χρόνια μας κοπανάνε αυτό το πράγμα ως δόγμα χωρίς ποτέ να έχει γίνει μια σοβαρή αξιολόγηση των δημοσίων πολιτικών και να έχουμε απτά αποτελέσματα ότι δίνουν και προωθούν αυτό που λέγεται ότι κάνουν. Επίσης, ισχυριζόμαστε ότι πιστεύουμε ότι οι διαφορετικές μεταρρυθμίσεις αγοράς εργασίας είναι προϋπόθεση για να αποκτήσει ανταγωνιστικότητα η οικονομία μας. Θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε διαμακρόν, αλλά δεν έχουμε χρόνο τώρα. Το μόνο που θέλω να πω είναι το εξή. Τι εννοούμε διαρθωτικές μεταρρυθμίσεις, γιατί όταν ε, εξετάζουμε τις συστάσεις, αυτές οι διαρθωτικές μεταρρυθμίσεις πηγαίνουν προς μία αποκλειστικά κατεύθυνση της μείωσης της κοινωνικής κάλυψης, της μείωσης της προστασίας στην αγορά εργασίας, υπέρ μιας θεωρητικής ανταγωνιστικότητας, η οποία ποτέ δεν αποδεικνύεται ότι υπάρχει. Να πω και ένα τρίτο και είναι ένα από τα παράδοξα της όλης προσπάθειας. Όταν αναλύουμε τις συστάσεις, μιλάνε πολύ για την βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας ή των συνταξιδοτικών συστημάτων, έτσι τα λέμε, το, τα συστήματα συλλογική διαπραγμάτευσης, τα μισθολογικά συστήματα. Και πού είναι το παράδοξο. Το παράδοξο είναι ότι η Ευρώπη αυτή τη στιγμή αρνείται να αναλάβει οποιαδήποτε αρμοδιότητα. Αλλά όταν πρόκειται για το ευρωπαϊκό εξάμεινο, έφνης εμφανίζονται αυτές οι αρμοδιότητες. Πιστεύω ότι πρέπει να σκεφτούμε. Υπάρχουν διάφορες απόψεις ε, επί του θέματος. Δεν είναι και το θέμα. Εγώ νομίζω ότι αυτό θα έχει επιπτώσει στους πολίτες πάντως, μεσοπρόθεσμα. Είναι περίπλοκο να λέμε ότι η Ευρώπη μπορεί να κάνει συστάσεις για τα συνταξιδοτικά συστήματα, αλλά όταν μιλάμε για θετικά πράγματα για τις συντάξεις, τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε από κοινού. Λέμε για συλλογικέ διαπραγματεύσει, ενώ θεωρούμε ότι δεν είναι κοινωτική αρμοδιότητα, έτσι. Για τα μισθολογικά, το ίδιο. Υπάρχει αυτό το παράδοξο. Και το τονίζω. Τρίτη παρατήρηση. Υπάρχουν πράγματα που εμφανίζονται λίγο ή ελάχιστα η ποιότητα της εργασίας. Δεν υπάρχει πουθενά, δεν εμφανίζεται. Δηλαδή, προωθείται η απασχόληση για την απασχόληση. Πάση θυσία. Αλλά ρωτήσαμε τους Ευρωπαίους για αυτή την απασχόληση, αυτού του απασχόληση. αυτά που συμβαίνουν σε ορισμένες χώρες, επί του προκειμένου, όπως η Γερμανία, είναι πολύ ενδιαφέροντα. Επίσης, από το 2008 και οι εργασίες σας το απέδειξαν, πάνω από 2 εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης καταστράφηκαν μέσω των λεγόμενων αναδιαρθρώσεων των επιχειρήσεων. Υπάρχουν ε, καθόλου συστάσεις για να βελτιώσουμε τη διαχείριση αυτή των ε, λεγόμενων ε, αναδιαρθρώσεων των επιχειρήσεων από πλευρά Κομισιόν. Ποτέ. Οι συστάσεις της ασχολούνται καθόλου με, την, με τα οικολογικά θέματα. Αν, αν αναλύσετε τις διάφορες συστάσεις προς τα κράτη-μέλη, δεν υπάρχει σχεδόν καμία αναφορά για τα περισσότερα κράτη-μέλη. Έχω άπειρα παραδείγματα που θα μπορούσα να δώσω. Αλλά θα τελειώσω γιατί ο χρονός είναι μετρημένος. Θέλω να κάνω τις εξής παρατηρήσεις τον αριθμό. Νομίζουμε ότι όλη αυτή η προσπάθεια γίνεται εκτός πλαισίου, χωρίς πλαίσιο. Λες και η κρίση δεν υπάρχει ή λες και την ξεχνάμε ή λες και υπάρχει μόνο σε επίπεδο δημοσίων α, λογαριασμών, δημοσιονομικού, στο δημοσιονομικό επίπεδο ας πούμε, πουθενά άλλου. Δεύτερο, όλη αυτή η προσπάθεια στέλνει ένα αρνητικό κοινωνικό μήνυμα στους περισσότερους Ευρωπαίους πολίτες και νομίζω ότι πρέπει σήμερα να θέσουμε το ερώτημα. Πρέπει να δώσουμε προκυκλικά ή αντικυκλικά μηνύματα σήμερα. Τι μηνύματα πρέπει να στείλουμε στους πολίτες. Πώς θα προετοιμάσουμε το μέλλον. Η κρίση που είναι το τρίτο. Δεν άλλαξε τίποτα. Νομίζω ότι δεν υπάρχει συντονισμός χωρίς όθηση. Η ο λόγος της Κομισιόν, ο κοινωνικός για την απασχόληση, είναι ακριβώς ο ίδιο. Ο ίδιος. Λες και η κρίση δεν άλλαξε τίποτα. Πώς μιλάμε σήμερα για ευέλιξη ασφάλεια σε ορισμένε χώρε, όταν δεν έχουμε τι ελάχιστε προποθέσει για αυτή την ευέλιξη ασφάλεια, ή ξεχάσαμε διάφορε φιλοδοξίε. Α πούμε, τη φιλοδοξία τη Κομισιόν που είχε για μια βαθιά μεταρρύθμιση των μηχανισμών των κοινωνικών δικαιωμάτων που χρειάζεται. Πώς θα προσαρμόσουμε τα κοινωνικά θέματα με την πραγματικότητα, ε, την πραγματικότητα των επιχειρήσεων, ε, τι καθεστώς έχουν οι εργαζόμενοι μέσα σε αυτές τις νέες επιχειρήσεις. Καμία παρατήρηση. Και τελευταία παρατήρηση. Μπορούμε να συντονίζουμε χωρίς να δώσουμε καμία, κανένα κίνητρο, καμία όφηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για αυτές, αυτά τα διαφωτιστικά σας σχόλια πολύ σημαντικά για την Επιτροπή μας, είτε μέσα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, είτε και εκτός. Όλες αυτές οι παρεμβάσεις εντάσσονται και στην δική μας πορεία. Ε, δημοσιονομική εξυγίανση δεν μπορεί να ε, είναι το μοναδικό εργαλείο αντιμετώπισης κρίσης, θα πρέπει να εξορροπηθεί. Αυτή είναι και η δική μας προσέγγιση και προσπαθούμε να βρούμε έναν τρόπο σήμερα το απόγευμα. Ανοίγω το ε, γύρο ερωταποκρίσεων, αν υπάρχουν ερωτήσεις θα θέσω εγώ την πρώτη. Στίβεν, κύριε Συγγήτρια, όχι, ο κύριος Σέρκας, ο κύριος Σέρκας. Θέλω να ευχαριστήσω τους ε, τέσσερις ε, φιλοξενούμενους μας ε, γιατί μας διευκρίνησαν μια πραγματικότητα αυτή που και εμείς αντιλαμβανόμαστε στην Επιτροπή μας. Η, κοινωνική οπτική γωνία δεν μπορεί να μείνει εκτός της διακυβέρνησης στην Ευρώπη. Η ευρωπαϊκή διακυβέρνηση είχε ως στόχο τη δημιουργία απασχόλησης, ε, την κοινωνική ένταξη, τη βελτίωση του βιωτικού επίπεδου. Και σιγά σιγά ε, γλιστρήσαμε, ολιστήσαμε προς ε, μια μονομερή αντιμετώπιση μέσω πολιτικών λιτότητας και αυτό που παλιότερα ήταν μέσο για την επιτεύξη στόχου έγινε αυτός σκοπός. Δηλαδή, οι στόχοι θα έπρεπε να είναι στην υπηρεσία των πολιτικών, όχι το αντίστροφο. Μάλλον, οι, υπηρεσίες, οι, πολιτικές θα έπρεπε να είναι στην υπηρεσία των στόχων και όχι το αντίστροφο. Είναι σαφές λοιπόν ότι κάτι πρέπει να αλλάξει και το είπαν οι τέσσερις ε, προσκεκλημένοι μας. Διότι τα πράγματα δεν χειροτερεύουν απλώς από την πλευρά των ε, πολιτών τα τελευταία χρόνια. Ακόμα και τα μακροοικονομικά αποτελέσματα χειροτερεύουν παρόλα τα όσα λέγονται. Δεν απογοητεύεται απλώς ε, ο πολίτης, ε, ε, διατρέχουν κίνδυνο τα ίδια τα συστήματά μας. Ορισμένα ερωτήματα που ήταν πολύ σημαντικά, πολύ κέρια. Γιατί δεν αξιολογούνται αυτές οι πολιτικές, γιατί οι πολιτικές ακολουθήθηκαν ε, από ψευδοεπιστημονικά ή επιστημονικοφανή δεδομένα. Όμως θα πρέπει να δούμε τα αποτελέσματα και με βάση αυτά να κρίνουμε τις πολιτικές. Κάτι τέτοιο δεν γίνεται. Αυτή τη στιγμή ή ακολουθείται μια δογματική προσέγγιση. Στην Ισπανία έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον εργαστήριο ιδεών και πριν από ένα χρόνο έγινε μια ε, διαρθρωτική μεταρρύθμιση η οποία εστιάστηκε αποκλειστικά στην αγορά εργασίας, δόθηκαν ενισχύσεις, εξασφαλίστηκε ευελιξία, ε, μειώθηκαν τα κόστη, ε, ελπίζοντας ότι δεν θα οδηγούμασταν σε ε, απολύσεις. Αντιθέτως, ότι θα οδηγούμασταν σε αύξηση της απασχόλησης. Πριν από ένα χρόνο έγιναν αυτά. Και η αλήθεια είναι ότι κατά τη διάρκεια αυτού του τελευταίου χρόνου αυτές οι μεταρρυθμίσεις όχι απλώς οδήγησαν σε μείωση, όχι δεν, οδήγησαν σε μείωση των ανέργων, αντιθέτως σε αύξησή τους. Και όχι μόνο δεν εξασφάλισαν την αύξηση των, ε, του αριθμού των ε, συμβάσεων αορίστου χρόνου, α, το ακριβώς αντίθετο αυξήθηκε ο αριθμός των προσωρινών συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Συνεπώ, η πραγματικότητα μα υπαγορεύει πω κάποιε αλλαγέ πρέπει να, κάνουμε. Γιατί αλλιώς κινδυνεύουμε να συγκρουστούμε με εμπόδιο. Ευχαριστώ. Δεν έχω να θέσω ερωτήματα. Θέλω να ευχαριστήσω του ομιλητέ μας για τους προβληματισμού του και να κάνω ένα προσωπικό σχόλιο απλώ. Άκουσα ότι η, κοινωνική, η οικονομική κρίση ε, και τα μέτρα λιτότητας είχαν επιπτώσεις στα, στις κοινωνικές πολιτικές και στην απασχόληση, με βαστά όσα είπαν οι ομιλητές μας. Άκουσα τα σχόλιά τους. Ο κύριος Τριόμφ μίλησε για αυτό το παράδοξο που υπάρχει στον προβληματισμό μας. Δηλαδή, δεν είμαστε πάντα συνεπείς ε, στη στάση μας και εξήγησε τι εννοούσε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συχνά συμμετέχει στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων μιας κρίσης μέσω της βοήθειας που δίνει σε μεγάλες επιχειρήσεις, ε, με βοήθεια προς τους εργαζόμενους, ε, αλλά εκ των προτέρων Όπω είπε κάποιος άλλος ομιλητή, δεν κάνουμε τίποτα. Έχουμε λίγα μέσα ω Ευρωπαϊκή Ένωση για να δράσουμε. Με κάποιε οδηγίε, ναι, με κάποιου προβληματισμού που δίνουμε δρούμε, αλλά δεν έχουμε πραγματική εξουσία να νομοθετήσουμε και να προβούμε σε διατάξει και να συντονίσουμε λόγω αυτή τη διαβόητη αρχή τη επικούρικότητα που θα πρέπει να αμφισβητηθεί. Νομίζω ότι έχουμε αρκετή ευελιξία σε αυτά τα πολιετή προγράμματα και σε αυτό το πολιτεσμο-συνομικό πλαίσιο ε, για να ασχοληθούμε με την απασχόληση. Θα πρέπει να κάνουμε ακριβώ τα ίδια, ε, να υπάρχει μια κοινωνική διακυβέρνηση ε, και στο κοινωνικό επίπεδο, αντίστοιχα με αυτά που κάναμε και τα οικονομικά θέματα. να, δούμε, να δούμε τα όρια της επικουρικότητας, να γίνει μια σχετική μελέτη για να δούμε τι περιθώρια έχουμε για το συντονισμό σε Ευρώπη. Και η πρόταση της Κομισιόν για την ασφάλιση της νεότητας, την εγγύηση για την νεότητα, πολύ ωραία ιδέα, αλλά και πάλι περνάει μέσα από τη βούληση των κρατών μελών. Πάντα εξαρτώματα από την βούληση των κρατών μελών. Δεν μπορούμε εμείς στο ευρωπαϊκό επίπεδο να προβληματιστούμε μαζί με το Συμβούλιο, μαζί με τα κράτη-μέλη, ούτως ώστε να υπάρξει καλύτερο συντονισμό. Το συμπέρασμα του κυρίου Τριόμφ είναι σωστό. Ε, μπορούμε να συντονίζουμε χωρίς να δίνουμε κίνητρα, χωρίς όθηση. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουμε περισσότερη ευκολία να έχουμε μια συνολική μακροοικονομική ας πούμε, θεώρηση ε, και έχουμε μια πιο συνολικότερη εικόνα του κοινωνικού τομέα. Αλλά ο, ο ρόλος μας δεν είναι απλώς να συντονίσουμε. Η μέθοδος του συντονισμού έχει δείξει τα όρια της, πόσο πεπερασμένη είναι, πόσο απαρχαιωμένη είναι. Νομίζω ότι τώρα θα πρέπει να υπάρξει σύγκληση πολύ πιο έντονη, σύγκληση λοιπόν, που με την διαφορετική αντιμετώπιση της επικουρικότητας θα επιτρέψει λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι πολύ πιο παρούσα στις κοινωνικές υποθέσεις ο Στίβεν Γιούγκ και η Έμιλι Τούρνεν. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστούμε και τους προσκεκλημένους μας σήμερα για τις ενδιαφέρουσες ιδέες και τις προκλητικές ιδέες που μας παρουσίασαν σε κάποιες ε, περιπτώσεις. Θέλω να κάνω κάποια συγκεκριμένα σχόλια και κάποια πιο ελληνικά. Μία συγκεκριμένη ερώτηση προς ε, τον Ζακ Τερπλά σε ό,τι αφορά το μηχανισμό για την ασφάλεια ανεργίας. Εξαιρετική ιδέα. Βλέπουμε όμως πόσο αργόστροφο είναι το Συμβούλιο σε όταν αφορά την ε, πρόθεση άλλων ιδεών και αυτό φαντάζομαι θα γίνει και με αυτή την ιδέα. Αναφερθήκατε προς το τέλος στο γιατί η Γερμανία ή η Ολλανδία θα προσυπέγραφαν την ιδέα αυτή. Δεν άκουσα ποια απάντηση δώσατε. Αν θα μπορούσατε να το αναπτύξετε αυτό, παρακαλώ. Δεύτερη συγκεκριμένη ερώτηση να συμφωνήσω μάλλον με τον ε, αυτό που είπε και ο κύριος Έρκας και ο κύριος Ντολπλά σε ό,τι αφορά τον τρόπο κατά τον οποίο οι NGS και τα διαφορετικά μεμοράντα κατανόησης που έχουν προσυπογραφεί με την Ιρλανδία και την Ελλάδα και την Πορτογαλία και την Ιρλανδία έχουν ε, εμπλακεί σε ό,τι αφορά τις ε, ρυθμίσει για τους ελάχιστους μισθού για τι συλλογικέ διαπραγματεύσει, γιατί δεν συμπεριλαμβάνονται τέτοια θέματα κοινωνικού κεφαλαίου στο, στις συνθήκες σε ό,τι αφορά την λιτότητα, ε, σε ό,τι αφορά τις εκθέσεις, τις αιτήσεις για τα κρατημέλη και τις εκθέσεις ανάπτυξης. Ε, να επανέλθω τώρα σε θέματα Είπατε ότι είναι απαραίτητη η λιτότητα, δεν είναι απαραίτητη και ότι είναι και λανθασμένη. Συμφωνώ από πλευράς ε, σοσιαλδημοκρατών, ε, όμως υποστηρίζουμε ότι ήταν απαραίτητη η δημοσιονομική πειθαρχία, αλλά διαφωνούμε με την ταχύτητα και το βάθος αυτής της ε, ε λιτότητες. Αναφερθήκατε και είπατε ότι θα πρέπει ο ιδιωτικός τομέας να δώσει ένα έναυσμα για να σπάσει ο κύκλος της ανεργίας. Συμφωνείτε ότι θα πρέπει να συμφωνήσουν και οι δημόσιες πολιτικές, να συμβάλλουν και οι δημόσιες πολιτικές σε ό,τι αφορά και την δημόσια ζήτηση. Γιατί αλλιώς πώς ε, θα δοθεί κίνητρο στον ιδιωτικό τομέα. Θα μείνει αβοήθητος ο ιδιωτικός τομέας και πώς θα προωθήσει την ανάπτυξη και τις θέσεις εργασίας. Νομίζω ότι θα πρέπει η δημόσιο, ο δημόσιος μακροοικονομικός τομέας να δώσει το κίνητρο και όχι ο ιδιωτικός τομέας. Συμφωνείτε με αυτά τα σχόλια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Εμιλή. Και μετά η κυρία Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να συνεχίσω στο ίδιο δρόμο που ε, στράφηκε και ο κύριος Χιούς. Θα πρέπει να γεφυρώσουμε κάποια άκρα. Αφενός, το ένα άκρο μπορεί κάπως να υπερβάλλουμε, αλλά στο ένα άκρο είναι η λιτότητα. Το όραμα ότι θα πρέπει να περιοριστεί, να συρρυκνωθεί ο δημόσιος τομέας, να συρρυκνωθεί ο μισθός και η κοινωνική προστασία. Και το άλλο άκρο είναι ότι θα πρέπει να υπάρχουν πολλές δαπάνες. Αυτά είναι τα δύο άκρα, χοντρικά και ότι θα πρέπει να γίνονται δαπάνες σε βάθος. Θεωρώ ότι αυτά τα δύο άκρα θα πρέπει να γεφυρωθούν σε μια τρίτη νέα θέση και νομίζω ότι η Επιτροπή μας ε, έχει τονίσει αυτή τη θέση σε όλες τις εκθέσεις και διακηρύττει ότι μια ισχυρή κοινωνία θα εξαρτάται από την στενή συνεργασία μεταξύ του δυτικού και του δημόσιου τομέα. Και εδώ σχολιάζω και αυτά που είπε η κυρία Αρκρέν. Είπατε ότι οι θέσει εργασία θα έρθουν από τον ιδιωτικό τομέα. Σύμφωνοι, αλλά ο ιδιωτικό τομέα εξαρτάται με τη σειρά του από τι ε, αποφάσει που λαμβάνονται σε επίπεδο τομέα. Θα ήθελα να τονίσω ότι στην παρούσα κατάσταση έχουμε μπει σε ένα φαύλο κύκλο. Οι επιχειρήσει, τα νοικοκυριά, όλοι ουσιαστικά δεν έχουν μια αισιοδοξία για το μέλλον και αυτό έχει παγώσει την οικονομία μας και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν έχουν παραλύσει επειδή είναι χαμηλή η ανάπτυξη. Είναι χαμηλή η ανάπτυξη, είναι χαμηλή η ζήτηση, γιατί όλοι φοβούνται το αύριο, γιατί ε, κόβουμε από τον ιδιωτικό τομέα και από το δημόσιο τομέα και αυξάνεται η ενεργεία. Και έτσι θεωρώ ότι βαθαίνουμε αυτή την κρίση και κάνουμε χειρότερο τον φαυλοκύκλο. Νομίζω ότι θα πρέπει να στραφούμε σε μια αισιοδοξία για την ανάπτυξη. Θα χρειαζόμαστε επενδύσεις. Σύμφωνοι. Δεν μπορούμε να κάνουμε επενδύσεις σε βάση νέων χρεών. Αυτό θα είναι πάρα πολύ δύσκολο σε πολλές, ε, στις πιο πολλές χώρες ε, της Ένωσης. Θα πρέπει να ε, υπάρχει δηλαδή χρηματοδότηση των επενδύσεων και το FTT αποτελεί μια άλλη πηγή επενδύσεων και χρειαζόμαστε καλύτερη συνεργασία, στρατηγικές ε, ε, εταιρικέ σχέσεις για νέες ε, θέσεις απασχόλησης, για την ενέργεια, για τις υποδομές. Αυτόν τον δρόμο πρέπει να τονίσουμε. Προς την κυρία Άλμγκρεκ, επειδή είστε από τη Σουηδία, εγώ την Δανία, ο Economist τόνισε ότι οι σκανδιναβικές χώρες ακριβώς αυτό κάνουν και γι' αυτό θεωρώ ότι οι επενδύσεις και η κοινωνική ασφάλεια μπορεί να υποστηρίζουν μακροπρόθεσμα και να συμβάλλουν μακροπρόθεσμα στην ανάπτυξη. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει αυτή η ισορροπία. Αυτή η Επιτροπή ουσιαστικά θεωρώ ότι γεφυρώνει αυτό το χάσμα, αυτά τα δύο άκρα, γιατί βρισκόμαστε σε μια πάρα πολύ επισφαλή κατάσταση σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Άρκιν, σας ευχαριστώ και καταρχάς να ζητήσω συγγνώμη γιατί άκουσα μόνο την τελευταία παρουσίαση. Σα ζητώ συγγνώμη, δεν μπόρεσα να έρθω πιο νωρί. Θα πρέπει να πω ότι συμφωνώ πάρα πολύ με αυτά που εξέφρασε η συνάδελφο Μιλτούνεν, ότι τίνουμε να κοιτάμε τα δύο άκρα. Ε, θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να βρούμε τη μέση εδώ. Μου έκανε εντύπωση αυτό που είπε ο τελευταίος ομιλητής, ότι κατά πόσον είμαστε προκυκλικοί στα μέτρα μας ή αντικυκλικοί. Μου φαίνεται ότι όλα τα μέτρα κινούνται προς μία κατεύθυνση και δεν υπάρχει εσωτερική ζήτηση σε πολλά κράτη-μέλη. Δεν υπάρχει δυνατότητα αύξησης των εξαγωγών, ίσως σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά όχι μέσα στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 0,6% συρρήκνωση της ευρωπαϊκής οικονομίας είναι πάρα πολύ ε, ανησυχητικό ποσοστό. Είναι τα πράγματα πάρα πολύ ανησυχητικά σε ό,τι αφορά τις ευρωπαϊκές οικονομίες και το κόστος, το δανεισμού είναι πολύ μεγαλύτερο. Άρα τα προβλήματα τα οποία ήδη υφίστανται επιτείνονται. Αυτό που θα ήθελα να γίνει και θέλω προς αυτή την κατεύθυνση να κάνετε προτάσεις, τι είδου αντικυκλικά μέτρα θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε και να ευχαριστήσω την Κάριτας γιατί κοίταξα την έκθεσή σας και είδα ότι αναφέρατε ειδικά την Ιρλανδία. Πολύ ωφέλιμο αυτό στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων άκουσα τον κύριο Τράγκη να μιλάει πριν από λίγε ημέρε για μια συμφωνία για το Ιρλανδικό Χρέο. και απάντησε σε έναν από του συναδέλφου μου, γιατί εγώ δεν μπόρεσα δυστυχώ να του θέσω ερώτηση, είπε ότι η κατάσταση στην Ιρλανδία είναι εξαιρετική. Ε, τυχερό ήταν που δεν κατάφερα να του θέσω ερωτήματα, γιατί τα στοιχεία τα έχουμε μπροστά μα και είναι απίστευτο ότι το λέει αυτό για μια τέτοια οικονομία, με τέτοιες ανάγκες. Απίστευτο. Ένα άλλο σχόλιο. Στη συζήτηση στο θέμα της ε, κυρίας ε, ε, Λόπος Μοντάνη το θέμα των πολλαπλασιαστών. Τι πιστεύετε, πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα. Κάποιοι μίλησαν για την ασφάλεια αυτή, την, για τους νέους, για την νεολαία. Ενδιαφέρουσα ιδέα. Πιστεύετε ότι θα πρέπει να υπάρχει και κάτι στη συνέχιση αυτού του μέτρου. Τι θα συμβεί στο μέλλον με όλο αυτόν τον κόσμο. Τελευταίο σχόλιο για να σχολιάσω και αυτά που είπε ο συνάδελφος και ο Στίβεν Χιούς. Χρειαζόμαστε διάφορες είδης και διάφορους ρυθμούς ε, δημοσιονομικής πειθαρχίας για, τα, για όλες τις χώρες σε ό,τι αφορά για παράδειγμα άλλα μέτρα που μπορούμε να λάβουμε για την ε, πάταξη της φοροδιαφυγής, για παράδειγμα, γιατί όλο ακούμε μέτρα λιτότητας να εξαγγείλονται. Μα πρέπει να βρούμε και άλλους μηχανισμούς για να βοηθήσουμε τις ευρωπαϊκές οικονομίες που βρίσκονται σε πολύ δύσκολη θέση. Ευχαριστώ. Θέλω και εγώ να πάρω το λόγο. Να πω δύο λόγια για το θέμα. Θα ήθελα να ρωτήσω τον Ζακ Τελπλά δύο πράγματα. Ε, μας είπε ότι οι ιδέες του δεν είναι καινούριε, παρόλο ότι είναι καινοτόμε. σε σχέση με την ε, ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την παράδοση. Όμως δεν μπορώ να φανταστώ ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να εφαρμοστεί χωρίς να θέσουμε το θέμα της, των όρων της κοινωνικής διαπραγμάτευσης. Όπως και στο, στην οικονομία, ο τετραγωνισμός του κύκλου είναι πώς είναι δυνατόν η εξυγίανση ε, να συνοδευτεί από διαφορετικές αλλαγές, παρόλο ότι πρέπει να ορίσουμε τελικά τι σημαίνει αυτό, ποιες είναι αυτές οι μεταρρυθμίσεις, έτσι και στον κοινωνικό τομέα τίθεται ένα παρόμοιο ερώτημα πολύ περισσότερο που σήμερα το πρωί το λέγαμε. Ο μακροοικονομικός διάλογος δεν, συν, δεν σε τίποτα, δεν χρησιμεύει. Τελικά η κεντρική τράπεζα μιλάμε τους κοινωνικούς εταίρους, απουσία μας. Βλέποντας όμως το τι συμβαίνει από πλευράς των κοινωνικών εταίρων, κάθε φορά που μιλάω με την Μπερναντέτ Σιγκολό ε, συζητάμε για την αυτονομία των κοινωνικών εταίρων στις ε, διαπραγματεύσεις. Εμείς αυτό το θεωρούμε απόλυτα απαραίτητο για το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο. Όμω, όταν βλέπουμε τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων και την ικανότητά του να διαπραγματευτούν, για παράδειγμα οδηγία μείωση του χρόνου εργασία, βλέπουμε ότι υπάρχουν προβλήματα στην αποτελεσματικότητα. Πώ θα τα συνδυάσουμε όλα αυτά. Και μετά, χρειαζόμαστε ένα εργαλείο που θα δίδει προσθέμενη αξία στο κοινωνικό τομέα και θα παίζει το ρόλο αυτόματου σταθεροποιητή ευρωπαϊκής διάστασης. Γιατί η δημοσιονομική εξυγίανση σε πολλά κράτη-μέλη οδηγεί σε καταστροφή αυτών των υπηρεσιών σταθεροποίηση σε εθνικό επίπεδο που υπήρχαν. Μήπως λοιπόν θα ήταν πιο εύκολο και πιο οικονομικό να υποστηρίξουμε ως πρώτο αυτόματο σταθεροποιητή την εγγύηση νεότητας. Δεν διαφωνώ με την ε, ασφάλιση ανεργίας, αλλά μήπως θα μπορούσαμε να βρούμε μια προσωρινή πρώτη λύση ως πρώτο βήμα. Γιατί τα 6 εκατομμύρια τα οποία δεσμεύτηκαν για την ε, εγγύης νεότητας ε, ήταν ένα καλό νέο και ίσως είναι πιο εφικτό να προωθηθεί αυτή η ιδέα καταρχήν. Δεύτερη ερώτηση για τον Κλοντ Μανουέλ Τριόμφ. Αφορά το εξή. Δεν συμφωνώ πλήρως με εσά που λέτε ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα. Είναι χειρότερα από πριν η κατάσταση. Έχει αλλάξει προς το χείρον. Μιλούσαμε με τον Ρόμπερτ Γκέμπελς πριν από λίγο και κάναμε πλάκα για το πώς οι κατευθυντήρες γραμμές διαφέρουν από την ε, πραγματικότητα. Πώς οι στόχοι δεν πετυχαίνονται. Μία από τις ανησυχίες μου είναι οι διαφορές ανάμεσα στο 121 και το 148 ε, που αφορούν την εξυγίανση και την απασχόληση, το οικονομικό και το κοινωνικό. Συνεπώς, αν κάτι πρέπει να δεχτούμε, είναι ότι θα πρέπει να κάνουμε κάτι μαζί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αλλά ποια είναι είναι οι προτεραιότητε στον κοινωνικό τομέα. Δεν ξέρω αν θέλει κανεί άλλο το λόγο. Ε, Τρώγοντα έρχεται η όρεξη, κύριε Μπενιό. Ένα σύντομο σχόλιο Γιατί δυσκολία στην οποία βρισκόμαστε. Είναι σαν ένα γυμνό δωμάτιο, να βρισκόμαστε σε ένα γυμνό δωμάτιο χωρίς εξόδους. Ε, υπάρχει μάλλον μόνο μία έξοδος με ένα μακρύ τούνελ. Ε, πολύ μακρύ και στο βάθος αχνά αχνά υπάρχει ένα φως, αμυδρό φως. Το πρόβλημα είναι ότι σε, υπό πιο συνήθεις ε, συνθήκες, σε τέτοια φάση θα αρχίζαμε να δημιουργούμε ε, ελλείμματα. Αλλά αυτό που συνέβη και ένας από τους χειρότερους μαθητές ε, ήταν το δικό μου κρατός είναι ότι ήδη είχαμε μεγάλα ελλείμματα σε περίοδο ευημερίας. Δηλαδή δεν έχουμε τώρα στη διάθεσή μας ένα ισχυρό μακροοικονομικό εργαλείο. Είχαμε δημιουργήσει δηλαδή ήδη ένα δύσκολο πρόβλημα από την περίοδο της ευημερία στην οποία βγαίνουμε. Και ο μόνος τρόπος για να προχωρήσουμε είναι μακροπρόθεσμες, διαρθωτικές, αλλαγές, όχι τόσο στην ποιότητα των δημοσίων δαπανών, αλλά στην, όχι στην ποσότητα, αλλά στην ποιότητα. Και θα πρέπει οι δημόσιες δαπάνες να πάνε σε εκείνους τους τομείς όπου θα εξασφαλίσουμε μια κάποια, ελπίζουμε, οικονομική ανάπτυξη. Για να κουνηθεί κάτι, να αλλάξει κάτι. Αλλά δεν είναι τίποτα το προφανές, δεν υπάρχει εύκολη διέξοδος, δεν υπάρχει εύκολη λύση. Δεν υπάρχει, α πούμε, το μαγικό ραβδάκι. Πρέπει να σταματήσουμε να ψάχνουμε τη μαγική λύση και να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε την ποιότητα των δαπανών και να μετακινήσουμε δαπάνες προς υποδομές, προς ε, έρευνα. Όσο γρηγορότερα το κάνουμε, τόσο καλύτερο. Αυτό δεν είναι ε, ερώτημα, είναι περισσότερο ένα σχόλιο. Δεν το απευθύνω προς κανέναν ειδικά, αλλά προς όλους. Σέργιο Γουτιέρες Πριώτο. Και συνεχεία κλείνω τον κατάλογο των ε, ομιλητών. Α, και μία κυρία, ο Σέργιο πρώτος. Gracias, Presidenta. Yo Ε, έχω μια αίσθηση έτσι απογοήτευσης αποκαρδιωτικό το πανόραμα. Βγάζουμε συμπεράσματα υπό το φως του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Στην τελευταία ολομέλεια του Στρασβούργου ε, θετήθηκε και μια έκθεση επιτροπής μας. Ταυτόχρονα όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο ε, κάνουν τα δικά τους μια πολιτική τελείως διαφορετική από αυτή που προτείνουμε εμείς. Σήμερα γίνεται η συζήτηση για την κατάσταση του, του κράτους στην Ισπανία και είναι κατά βάση ένα κράτος απελπισίας. Εδώ και τρία χρόνια ακολουθούμε την στρατηγική η οποία μας επιβάλλεται από το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και, την, και από την πολιτική μακροοικονομικού συντονισμού και αυτό που έχουμε καταφέρει είναι περισσότερη φτώχεια, μικρότερη ανάπτυξη και περισσότερο ευρωσκεπτικισμό διότι και από πολιτική σε πλευράς πρέπει να διαρωτηθούμε αυτή η πολιτική που μας υπαγορεύεται ε, εξ αρχής, ε, αυτή η σιδηρά πειθαρχία, δημοσιονομική πειθαρχία, ε, τι, δημιουργεί, τι αποτελέσματα δίνει. Δίνει, προκαλεί ένα πραγματικό ευρωσκεπτικισμό, ε, εμπνέει δυσπιστία. Οπότε η ερώτηση είναι εξή από τις συστάσεις που απευθύνει η Επιτροπή κάθε χρόνο στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Ε, αυτές, κάποια από αυτές τις στάσεις όλες μας οδηγούν σε καλύτερη κατάσταση, μας οδηγούν σε βελτίωση. Η απάντηση είναι όχι. Όλο αποτυγχάνουμε ε, στην εκπλήρωση των στόχων μας. Έτσι κι αλλιώς ε, δεν παρακολουθούμε τους κοινωνικούς στόχους, δεν μετρούμε ούτε αξιολογούμε το αν ε, επιτυγχάνονται, αλλά και σε οικονομικό, καθαρά οικονομικό επίπεδο αποτυγχάνουμε. Συνεπώς δεν είμαστε αρκετά χειρότερα από πέρσι, είμαστε αρκετά χειρότερα από ό,τι ήμασταν πριν από μία εβδομάδα. Ακόμα και η συμφωνία για τον προϋπολογισμό ε, που επήλθε είναι πολύ χειρότερη από αυτό που ζητούμε εμείς ως Επιτροπή. Συνεπώς, ε, η προσπάθειες που κάνουμε σε εθνικό επίπεδο θα έπρεπε να συνοδεύονται από μια τουλάχιστον συμφωνία για τον προβλησμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα έδινε ευκαιρίες ανάπτυξης. Όχι, το αντίθετο. Χρειαζόμασταν συγκεκριμένες παρεμβάσεις για την οικονομική ανάπτυξη. Και ταυτόχρονα Ενώ συζητούμε το δίλημα ανάπτυξη ή λιτότητα, συζητώντας με τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, μας ε, λέγεται ότι ε, μας αναφέρθηκε ότι οποιαδήποτε απόκληση από τη λιτότητα θα δημιουργούσε αμφιβολίες για τη δυνατότητα της επιβίωσης του ευρώ. Ε, Ε, πολλοί μιλούν για το ότι, πολλοί πολιτικοί ενώ μιλούν, λένε ότι δεν θα πρέπει να αμφισβητηθεί το ευρώ, αλλά κανένας δεν λέει ότι δεν θα πρέπει να αμφισβητηθεί το κοινωνικό μας μοντέλο. Και πρέπει να έχουμε πάντοτε στο μυαλό μας και τελειώνω με αυτό. Ε, να, να πω ότι μου άρεσε η παρέμβαση του εκπροσώπου της για αυτό το θέμα. Θα πρέπει να εξετάζουμε πάντοτε ε, τον κοινωνικό αντίκτυπο των μέτρων και των πολιτικών που υπαγορεύει το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Μα λένε, μα υπόσχονται αύξηση τη ανταγωνιστικότητα. Και εγώ διερωτώ, με ποια είναι αυτή η ανταγωνιστικότητα που μα υπόσχονται μέσω μεταρρυθμίσεων, ε, σιακών μεταρρυθμίσεων που ε, κάνουν πιο φτωχούς τους πελάτες, τους πολίτες ε, και μην ξεχνάμε ότι μεταξύ των πιο ανταγωνιστικών χωρών καμία από τις πέντε πρώτες δεν χαρακτηρίζεται από ε, ε έλλειψη προστασίας ε, των εργαζομένων, από ε, προσωρινές θέσεις εργασίας κλπ. Συνεπώς, ακολουθούμε ένα λάθος δρόμο και μας ε, ε, οδηγούν σε ένα σημείο που σε, λίγα καιρό, σε λίγο καιρό δεν θα αναγνωρίζουμε πλέον το κοινωνικό μοντέλο που χτίζαμε εδώ και 30 χρόνια. Ε, Εγώ έδωσα το κακό παράδειγμα και εσείς συνεχίσατε προς την ίδια κατεύθυνση. Κυρία Φοντανιέ, δεν θα απαντήσω στον συνάδελφο από ε, την Ισπανία. Δεν θα μιλήσω για την πολιτική της Ισπανικής κυβέρνησης τον τελευταίο καιρό. Δεν είναι το πιο κατάλληλο πλαίσιο. Ε, δεν θα μιλήσω ε, για απελπισία αλλά για ελπίδα. Νομίζω ότι τα πράγματα γίνονται σωστά στην Ισπανία. Και θα δούμε τα αποτελέσματα σύντομα. Η εργασιακή η μεταρρύθμιση, οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις γενικότερα δεν δίνουν αποτελέσματα σε ένα χρόνο. δεν θα μιλήσω για αυτό το ζήτημα. Οι παρεμβάσεις των ε, προσκεκλημένων μα ήταν πολύ ενδιαφέρουσε. Συμφωνούμε νομίζω όλοι ότι χρειαζόμαστε ε, εξισορρόπηση ε, του προπολογισμού για να εξασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα του κοινωνικού μας συστήματος. Όμως η λιτότητα δεν μπορεί να υποσκάψει την ανάπτυξη για το μέλλον. Ε, να σας πω την εξή σκέψη. Μιλάμε πολύ για το πώς μπορούμε να βγούμε από την κρίση, πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε απασχόληση, πώς είναι δυνατόν να βοηθήσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μέτρα δηλαδή που είναι κυρίως μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα και μετά ο εκπρόσωπο τη Κάριτα μα ε, μίλησε για το καθαρά βραχυπρόθεσμο, για τα βραχυπρόθεσμα μέτρα, για το τώρα, ε, το παρόν που επήγει, γιατί ε, για την σημερινή φτώχεια δεν μπορούμε να μιλάμε με μέτρα του αύριο ή του μεθαύριο. Συνεπώ υπάρχουν δύο διαφορετικέ οπτικέ γωνίε και θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη και να στείλουμε αυτό το μήνυμα στο Συμβούλιο. Πρέπει να γίνουν μεταρρυθμίσεις, αλλά θα πρέπει να ληφθούν και άμεσα μέτρα. Και αυτό είναι το συμπέρασμα το οποίο θα έβγαζα εγώ από την σημερινή ακρόση. Ευχαριστώ. Αν συμφωνείτε θα δώσω ξανά το λόγο στους προσκεκλημένους μας με την ίδια σειρά, ξεκινώντας από τον Ζακ Δελπλά. Παρακαλώ πολύ περιοριστείτε στα πέντε λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Για τη συζήτηση περί λιτότητας. Η συζήτηση που ξεκίνησε από τον Ολιβιέ Μπλονσάχ αφορά την Γερμανία, τις κατοχώρες στη Γαλλία, αλλά επουδενή τις χώρες του Νότου. Ε, στις χώρες του Νότου ε, δεν υπάρχει θέμα λιτότητας, διότι κανείς δεν θα τους δάνειζε έτσι κι αλλιώς. Το πρόβλημα της ε, Ισπανίας είναι ότι οι κυβερνήσεις Αθηνών και Θαπατέρο επέτρεψαν μια φούσκα του κατασκευαστικού τομέα, η οποία εξεράγει. Η ανεργία της Ισπανίας δεν είναι κυκλικό φαινόμενο, ε, είναι πρόβλημα ότι, το πρόβλημα προέρχεται από το ότι υπήρχαν πολλοί που κατασκεύαζαν σπίτια. Ακίνητα. Δεύτερον, μου έκανε μία ερώτηση ο Γερμανός, ο Άγγλος συνάδελφος, γιατί θα συμμετείχαν σε ένα μηχανισμό ασφάλισης ανεργίας η Γερμανία και η Ολλανδία. Η εύκολη απάντηση είναι για το μακροπρόθεσμο πλαίσιο. Δεν θέλω να επισέλθω σε λεπτομέρειες, αλλά δίνουμε ασφάλεια για την κυκλική ανεργία και χρηματοδοτούμε την ε, ε, διαφορά μεταξύ της ε, ανεργίας αυτής και της κύκλικής ανεργίας είναι, επειδή κοιτάμε δηλαδή μόνο την κυκλική ανεργία, το ποσό είναι ουδέτερο. Σε 5-7 έως 7 χρόνια η Γερμανία θα είναι καθαρός αποδοχέας τέτοιων κονδυλίων. Είναι δηλαδή ουδέτερο τελικά, ούτε αρνητικό ούτε θετικό το αποτέλεσμα για όλες τις χώρες. Μία άλλη πιο δύσκολη ε, απάντηση είναι Όπως είπε και ο Ισπανός συνάδελφός σας, η Ισπανία είναι μια ορολογική βόμβα σε ό,τι αφορά την ανεργία. Στο σύνολό της δεν μπορούμε να έχουμε 25 έως 30% ανεργία στο Νότο, ιδιαίτερα στην Ισπανία που είναι μεγάλη χώρα. Και έτσι απαντάω την ερώτησή σας. Ε, είπατε τι καλός που είστε, αλλά να σας πω ότι έκανα μια πρόταση Blue πριν από 3-5 χρόνια. Όλοι μου είπαν ότι είσαι τρελός. Δεν έχει εφαρμοστεί, αλλά έχει κατατεθεί. Ο όλεθρος ε, ως προς την ανεργία. Αν δεν επιλύσουμε το θέμα της ανεργίας, αν δεν πέσει η ανεργία στην Ισπανία, στην Ελλάδα, στην Πορτογαλία, θα υπάρξει έκρηξη. Η ε, Ισπανία θα πτωχεύσει, ενδεχομένω να αναγκαστεί να φύγει από το ευρώ. Ακόμα και αν όλα τα κόμματα είναι υπέρ της ε, Ευρώπης. Ο λόγος λοιπόν που η Γερμανία ε, κάνει ό,τι κάνει είναι ότι θέλει να αποφύγει μία προς τα έσω ε, ρήξη και καλά κάνει. Και δεν θα το αποτρέψουμε αυτό αν δεν, απευθύνουμε, αν δεν απαντήσουμε στο ερώτημα στο θέμα της ανεργίας. Και οι βορειοσκήνωτες χώρες και τα βασικά μέρη, θέλουμε να έχουμε ασφάλεια, θέλουμε να έχουμε μέτρα τα οποία μπορούν να επιψηφιστούν από όλα τα κόμματα του πολιτικού φάσματος. Δεν θέλουμε κάτι υπερβολικά πολλωμένο. Κυρία Πρόεδρε, για να απαντήσω στα δικά σας ερωτήματα. Ε, κοινωνική διαπραγμάτευση. Εγώ είμαι οικονομολόγος. Ε, αλλά δεν μπορούμε να έχουμε την αυταπάτη ότι μόνο η κοινωνική εταίρεια είναι αυτόνομη. Γιατί, γιατί η Ευρώπη χαρακτηρίζεται από πολύ διαφορετικά κοινωνικά συστήματα και στην ε, πρότασή μας ε, πρέπει τα κράτη να δεχτούν ε, να καταβάλουν πληρωμές που θα είναι δημοσιονομικής φύσεως. Συνεπώς, οι κοινωνικοί εταίροι πρέπει να έχουν ρόλο, είναι θεμητό, αλλά δεν θα είναι δυνατόν μόνοι τους να αποφασίσουν ε, την κατανομή και την δέσμευση ε, δημοσιονομικών ποσών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνεπώς, χρειάζεται μια συμφωνία ανάμεσα στις πολιτικές αρχές, την εκτελεστική εξουσία, ε, το κοινοβούλιο και τους κοινωνικούς εταίρους. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν θα ήταν δυνατό να φανταστούμε ότι οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι στις Βρυξέλλες θα αποφάσιζαν το, τη μορφή που θα, η, θα πάρει η Ευρωπαϊκή Ασφάλιση Ανεργίας. Όποια μορφή και να πάρει αυτή. Αν μπορούμε να προβλέψουμε έναν σταθεροποιητή για τους νέους. Νομίζω ότι όσα γίνονται για τους νέους είναι πολύ καλά. Ε, πρόκειται για μια διαρθρωτική πολιτική, όχι κύκλικης φύσεως. Εμείς έχουμε μιλήσει για το Erasmus Eco. Το Eco δεν είναι από το οικονομία, αλλά για τον Umber, από τον Umberto Eco. Umberto Eco πριν από ένα χρόνο παρουσίασε την εξή ιδέα, το καλύτερο, ότι το καλύτερο ευρωπαϊκό πρόγραμμα είναι το Erasmus. Ε, όμως το έρασμος αφορά αυτούς που πιστεύουν στην Ευρώπη ε, και μπορούν να μετακινηθούν. Όμως χρειάζονται έρασμος και για πολλά άλλα επαγγέλματα, ταξιτζίδες, υδραυλικούς κλπ. Οπότε η ιδέα του Ουμπέρτο Έκο ήταν το έρασμος να γίνει πραγματική πλατφόρμα κινητικότητα στην Ευρώπη. Όχι μόνο για τους ε, φοιτητέ. Αυτό προτείνω. Να πάρουμε χρήματα από, τον, από τα διορθωτικά ταμεία και να τα επενδύσουμε σε ένα διευρυμένο έρασμο, το οποίο εγώ θα το ονόμαζα έρασμο Σουμπέρτο Έκο. Και κάτι άλλο. Αν δεν έχουμε ιδέες για τη μείωση του ποσοστού ανεργίας, δεν πρόκειται να έχουμε μέλλον, να εξασφαλίσουμε μέλλον και για το ευρώ. Η συζήτηση για τους πολλαπλασιαστές δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Η ανεργία της Ισπανίας είναι κυρίως διαρθρωτική. Υπάρχει ένα εκατομμύριο άτομα τα οποία ε, δούλευαν στον κατασκευαστικό τομέα και τώρα πια δεν δουλεύουν εκεί. Δεν είναι θέμα κυκλικό. Τι θα κάνουμε με αυτού, πώ μπορούμε να μεταρρυθμίσουμε την αγορά εργασία στην Ισπανία. Αυτή τη στιγμή η Ισπανία έχει τη χειρότερη αγορά εργασία στην, στην Ευρώπη. Πώ μπορούμε να τη βοηθήσουμε να μεταρρυθμίσει την αγορά εργασία τη. Ε, Ευχαριστώ. Η κυρία θα μιλήσει. Ευχαριστώ. Η Ευρώπη αντιμετωπίζει μια τεράστια πρόκληση. Θα πρέπει να μειώσουμε την ενεργεία. Θα πρέπει να αυξήσουμε την απασχόληση. Συμφωνήσαμε ότι ο δημόσιο τομέα ασφαλώ θα πρέπει να κάνει επενδύσεις και να παρέχει υπηρεσίες, αλλά θα πρέπει να είναι και αποτελεσματικό, αποδοτικός. Οι προτεραιότητε θα πρέπει να είναι στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της έρευνας και της καινοτομία. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις παρέχουν 60 έως 70% των θέσεων απασχόλησης στην αγορά. Πίσω από κάθε μικρομεσαία επιχείρηση έχουμε ένα άτομο που μπορεί να πάει στην ε, τράπεζα για δάνειο. Στην Σουηδία βλέπουμε ότι πληρώνουμε 3% παραπάνω επιτόκια από ότι μεγάλες επιχειρήσεις. Υπάρχουν διοικητικά άχτη τα οποία δεν περιορίζονται Κατά 25% όπως ακούσαμε ότι έχει τεθεί στόχος σχετικό. βλέπουμε ότι αυξάνεται το γραφειοκρατικό άχθος αντιθέτως. Άρα μας δεσμεύουν τα γραφεία και δεν προσανατολιζόμαστε στις πωλήσει. Θα πρέπει να ενθαρρύνουμε τα άτομα να, ξεκινούν, να ξεκινούν επιχειρήσεις και να τις αναπτύσσουν για να δημιουργούν θέσεις απασχόλησης. Επίσης συμφωνούμε ότι υπάρχει έλλειψη πίστης για το μέλλον. Και αυτό συνδυάζεται με τα άτομα, με τους ιδιώτες. Θέλουμε να δημιουργούν θέσεις εργασίας, αλλά θέλουμε και δίκαιες ρυθμίσεις. Χρειαζόμαστε σε εθνικό επίπεδο να εφαρμοστούν οι νομοθεσίες για τις μικρές επιχειρήσεις. Να σκεφτόμαστε από το χαμηλό επίπεδο για να αυξήσουμε το ποσοστό απασχόλησης. Ευχαριστώ. Ο Γιώργεν Νούνιεθ Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να επικεντρωθώ στο ερώτημα του τι θα ακολουθήσει αυτό το πρόγραμμα εγγύησης ασφάλισης ε, της νεολαίας. Στην ε, Κάριτα έχουμε καλές ε, εμπειρίες από την Ισπανία, από τη Γερμανία, όπου ο διάλογος μεταξύ δημοσίου τομέα και ιδιωτικού τομέα και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων δηλαδή βασικά, αλλά και με τους παρόχους ε, δημοσίων κοινοφελών ε, υπηρεσιών όπως η Κάριτας, δημιουργούν ε, θέσεις εργασίας στον τομέα της φροντίδας ε, της, ε, των πράσινων θέσεων εργασίας ε, στον τομέα της κοινωνική οικονομίας, όπου θεωρούμε ότι θα πρέπει να προσανατολιστούν και οι μελλοντικές πολιτικές. Υπάρχουν δηλαδή δυνατότητες, υπάρχουν εμπειρίες, αλλά θα πρέπει να υπάρχει ένας συντονισμό προκειμένου να στεφτεί με επιτυχία για όλη την Ευρώπη αυτό το ζήτημα και όχι μόνο για τους λίγους εκλεκτούς. Ευχαριστώ. Ο κύριος, Ο κύριος Μπορώ να συνοψίσω την απάντησή μου προς όλες τις ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις που μου έγιναν συνοψίζονται ως εξής. Πώς μπορούμε να προχωρήσουμε σε απαντήσεις όχι κυκλικές αλλά αντικυκλικές στον κοινωνικό τομέα. Η απάντηση μου δεν είναι μονοσήμαντη. Το μόνο που θέλω να πω είναι το εξή. Και πριν από την κρίση, αλλά και η κρίση και το ευρωπαϊκό εξάμεινο δείχνουν ότι η κοινωνική προσέγγιση της Ευρώπης έχει φτάσει στο τέλος ζωής της. Δεν καταλάβαμε, δεν συνειδητοποίησαμε τη διάσταση των πραγματικών μεταρρυθμίσεων που έγιναν και στον παραγωγικό ιστό μας και στο μισθολογικό ιστό μας. Πρέπει να βρούμε κάτι καινούριο, μια νέα προσέγγιση. Ίσως είναι αβάσταχτο αυτό σήμερα. Αυτό που είναι αβάσταχτο ε, είναι ότι ακούμε τα ίδια μπλα μπλα που ακούμε εδώ και 10 χρόνια με την ίδια σοβαροφάνεια από τα ίδια θεσμικά όργανα ενώ αυτές οι απόψεις, αυτές οι προσεγγίσεις δεν έχουν δώσει αποτελέσματα. Το θέμα δεν είναι αν είμαστε υπέρ ή κατά. Το θέμα είναι ότι αυτά δοκιμάστηκαν και απέτυχαν. Επομένως, τι μας, μένει, μας μένουν δύο στοιχεία. Την έννοια της κοινωνικής καινοτομίας πρέπει να την αντιμετωπίσουμε. Δεν μπορούμε να το γλιτώσουμε αυτό. Πολλοί μίλησαν για το θέμα της αυτονομίας. Και εσείς, Πρόεδρε, και τα λοιπά. Και πολλοί ομιλητές. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να μιλάμε για αυτονομία του κοινωνικού διαλόγου και να βάζουμε τελεία εκεί. Ούτε μπορούμε να πούμε ότι μια και δεν ε, λειτουργεί, ε, οι δημόσιες αρχές θα πρέπει να αναλάβουν αυτές ε, και να παίξουν το ρόλο τους, μια και δεν λειτουργεί ο διάλογος. Ε, το θέμα είναι να πούμε σήμερα ο αυριανός κοινωνικός διάλογος, από τι θα αποτελείται εκπλήσωμε που σήμερα έχουμε ε, αυτές τις έννοιες της κοινωνικής ευθύνης, της επιχείρησης, της, του ανοίγματο σε όλους τους συμμετέχοντες, αλλά όταν κοιτάμε τον κοινωνικό διάλογο, πώς λαμβάνει η χώρα σήμερα, ο κοινωνικός διάλογος είναι κλειστός, δεν είναι ανοιχτός στους νέους συμμετέχοντες. Πρέπει να κάνουμε μια προσπάθεια καινοτομίας. Θα σας, κάνω, θα σας δώσω ένα τελευταίο παράδειγμα στο θέμα ε, που αφορά την απασχολησιμότητα, έτσι. Τελευταίο, σας διαβεβαιώ. Επί χρόνια, νομίζω, ότι λέγαμε ότι τα παθητικά μέτρα δεν αρκούν, χρειάζονται ενεργητικά μέτρα. Είναι όμως δύο παράλληλα πράγματα, παράλληλα κανάλια που δεν λειτουργούν από κοινού. Πώς θα τα, θα κάνουμε αυτά ένα συνεκτικό πακέτο. Θα, δώσω ένα παράδειγμα. Αφενός για τους ανέργους και αφετέρου για τους ε, εργαζόμενους πιστεύω και μπορώ να σας σοκάρει ότι σε μια Ευρώπη στην κρίση δεν μπορούμε να γλιτώσουμε ένα νέο προβληματισμό για μια κάποια κάποια μορφή μείωση του χρόνου εργασία. Γιατί? Γιατί έχει μειωθεί ούτω ή άλλω ο χρόνο εργασία. Το θέμα είναι πώ μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε έξυπνα αυτή τη μείωση. Για να δώσουμε άδειε, όχι. Πώ θα συνδυάσουμε σήμερα τον μειωμένο χρόνο εργασία θα τον μοιράσουμε πιο δίκαια, ούτω ώστε να εξυπηρετήσει την απασχολησιμότητα του αύριο. Εδώ πρέπει να σκεφτούμε διάφορα πράγματα, ούτω ώστε ε, να επιτρέψουμε οι πιο ευπαθεί εργαζόμενοι να μειώσουν το χρόνο εργασία του μεν, αλλά να εξασφαλίσουμε μεγαλύτερη απασχολησιμότητα για αυτού αύριο. Αυτέ είναι κάποιε ιδέε που ρίχνω στο τραπέζι. Δεν θα υπάρξει ε, συντονισμό χωρί κίνητρα, δεν θα υπάρξουν κίνητρα χωρί καινοτομία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τους τέσσερις ομιλητές μας για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα ακρόαση. Νομίζω ότι υπάρχουν πράγματα που θα εξελιχθούν και νομίζω ότι όλα όσα ακούστηκαν ήταν πολύ ενδιαφέροντα για τους συναδέλφους. Μην ξεχνάμε ότι αυτά τα θέματα πολύ γρήγορα θα ξαναείνει στο προσκήνιο. Εν ώψη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Ιουνίου. Τελειώσαμε λοιπόν με την ακρόαση αυτή. Ευχαριστώ τους εμπειρογνώμονες. Και πάμε στο σημείο 15 της ημερησίας διάταξης. Θα δώσω το λόγο στην κυρία McIntyre για το σχέδιο γνωμοδότησης για την Επιτροπή Περιβάλλοντος, για τους βασικούς κανόνες ασφαλείας, για την υγειονομική προστασία από τους ε, κινδύνους που προκύπτουν από την έκθεση σε ιονίζουσες ακτινοβολίες. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ. Αυτό το σχέδιο οδηγία για τι ιονίζουσε ακτινοβολίε. σκοπό έχει να απλοποιήσει τις υφιστάμενες ρυθμίσει και ε, να συνενώσει τις πέντε υφιστάμενες οδηγίες σε μια νέα οδηγία για τα πρώτα ασφαλείας και σκοπό έχει να ενσωματώσουν τις τελευταίες συστάσεις της Διεθνούς Επιτροπής για την Ραδιολογική Προστασία, την ICRP όπως ονομάζεται, και να εναρμονίσει το ευρωπαϊκό καθεστώς με τα βασικά πρότυπα ασφαλείας της Διεθνούς ε, Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας. Είναι σημαντικό η χρήση ιονίζους ε, ακτινοβολίας ε, είναι σημαντικό θέμα για πολλές βιομηχανίες που αποτελούν και βασική πηγή θέσεων απασχόλησης και γι' αυτό τα, τα πρότυπα για την ε, προστασία των εργαζομένων έχουν τεθεί από το 59. Εγώ υποστηρίζω την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μια πιο συνεκτική προσέγγιση και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να κοιτάξουμε μια προσέγγιση βάσει επιστημονικών τεκμηριωμένων στοιχείων. όπω ε, θα θυμάστε ίσως και όχι, το αρχικό χρονοδιάγραμμα για την γνωμοδότηση αυτή ήταν πάρα πολύ ε, γρήγορο. Γι' αυτό λοιπόν κατέθεσα πολύ λίγε τροπολογίε, Ωστόσο, μετά από τι περαιτέρω ε, διαβουλεύσεις με τους εμπειρογνώμονες, αναθεώρησα κάποιε από τι τροπολογίε μου για να συμπεριλάβω νέα επιστημονικά στοιχεία τα οποία ανέκυψαν στο μεταξύ. Η έκθεση αυτή είναι σε συνεργασία με την Επιτροπή Περιβάλλοντος. Υπάρχουν κάποιοι τομείς όπου έχουμε κοινή αρμοδιότητα και σε κάποιους άλλους τομείς έχουμε αποκλειστική αρμοδιότητα. Είναι σημαντικό παρ' όλα αυτά να κοιτάμε εμείς πιο πολύ τα θέματα απασχόλησης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα μέλη της Επιτροπής που κατέθεσαν τροπολογίες. Ελπίζω να συνεχίσουμε την καλή συνεργασία με όλες τις ομάδες προκειμένου να καταλήξουμε σε μια καλή ισορροπημένη γνωμοδότηση προς την Επιτροπή ΕΝΒΗ. Σύντομα θα διοργανώσω συνεδρίαση των κοιοδών εισηγητών για να συζητήσουμε κάποιες λεπτομέρειες και κάποιες ε, στοιχεία θα πρέπει να τα κοιτάξουμε ιδιαίτερως. Δύο θέματα ενδεχομένω να παρουσιάσουν ε, αμφισβητήσεις. Το θέμα πρώτο είναι τι θα γίνει με τα άτομα κάτω των 18. Εγώ θα αποσύρω τη δική μου τροπολογία υπαριθμών 7 για το άρθρο 12 που έχει να κάνει με τα άτομα 16 έως 18 ετών. Με έπεισαν ότι δεν είναι σωστή η τροπολογία που κατέθεσα, αλλά θα πρέπει να κοιτάξουμε. Νομίζω ότι και ο κύριος Όρη έχει καταθέσει σχετικές τροπολογίες και η κυρία Στάινμπρουκ και άλλοι που είναι αντιφατικές. Άρα θα πρέπει να κάτσουμε και να βρούμε έναν λογικό συμβιβασμό. Θεωρώ ότι το πιο αμφιλεγόμενο θέμα. Οι πιο αμφιλεγόμενε τροπολογίε είναι εκείνες που θέλουν να συμπεριλάβουν και του, τα άτομα που ταξιδεύουν συχνά με αεροπλάνο, τους frequent flyers. Νομίζω ότι αυτό θα καλύπτει κάθε βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καταρχά. Δεν έχω πιστεί ακόμα με ακλόντα επιστημονικά στοιχεία για να υποστηρίξω αυτή τη θέση. Ξέρω ότι δεν είναι εδώ πέρα η συνάδελφος και ξέρω ότι η κυρία Στάνερα, αλλά που έχει πάρα πολύ... είναι πολύ πεπισμένη ότι θα πρέπει να συμπεριληφθεί αυτή η κατηγορία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ελπίζω να καταφέρουμε να κάνουμε κάποιους συμβιβασμούς με τους κοιόδης ε, εισηγητές και να υποβάλουμε καλές προτάσεις προς την Επιτροπή. Να σας ευχαριστήσω λοιπόν και πάλι συνάδελφοι και να ακούσω τα σχόλιά σας αν έχετε ενδεχομένω. Ευχαριστώ ο κύριος ε, Όρη και μετά ο κύριος Μπενιών. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την καλή δουλειά της. Ευχαριστώ κύριε Μακιντάιρ. Είπαμε ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα θέματα απασχόλησης στον τομέα αυτό. Ε, έτσι μας είπαν. Εγώ δεν συμφωνώ. Υπάρχει και μια άλλη ευρωπαϊκή αρμοδιότητα, η υγεία και η ασφάλεια στον χώρο εργασία. Και νομίζω ότι είμαστε υπεύθυνοι και για αυτό το τομέα. Άρα λογικό είναι να εργαστούμε και από αυτού του θέματος και νομίζω ότι υπάρχει και εντολή. Ε, έχουμε απόλυτα το δικαίωμα να δώσουμε τη γνώμη μας και για αυτό το θέμα. Στη γνωμοδότηση και στις τροπολογίες προκύπτει ότι ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε τα θέματα, αυτή την ισορροπία που ψάχνουμε, ότι είναι κοινό στην Ευρώπη, να το κάνουμε με τον ίδιο τρόπο σε όλη την Ευρώπη, από τη μία και από την άλλη, ποιε είναι οι αποκλήσει σε εθνικό επίπεδο από αυτή την κοινή γραμμή, και το πώς θα εξορροπήσουμε τα δύο. Η κυρία Μακεντάρη είπε ότι θα πρέπει να εναρμονίσουμε πολύ τους κανόνες. Αυτό βγαίνει ξεκάθαρα από την έκθεση, αλλά εγώ πιστεύω ότι αυτό θα ήταν η σωστή προσέγγιση. Το λέω για λόγους υγείας και ασφάλειας. Στο κάτω-κάτω μιλάμε για ανθρώπινες ζωές και για την ανθρώπινη υγεία. Και όταν μιλάμε για τέτοια θέματα, λογικό είναι να έχουμε απόλυτα ενιαίους κανόνες. Και έχω και μια άλλη άποψη που αφορά, που βασίζεται μάλλον στον ανταγωνισμό ανταγωνιστικότητα. Ε, ούτως ή άλλως μιλάμε για διαφορετικές συνθήκες, ε, εργασιακές σχέσεις, συνθήκε στι οποίε δραστηριοποιούνται επιχειρήσει, και θα πρέπει όλοι όσοι συμμετέχουν στον ανταγωνισμό στην αγορά να συμμετέχουν επίσης όρει. Ε, οι τροπολογίες μου ε, βασικά απορρέουν από αυτά που σας είπα ήδη. Μερικές φορές πιστεύω όμως ότι οι προϋποθέσεις το παρακάνουν Ίσως είναι υπερβολικό να ζητήσουμε ορισμένα από αυτά τα σημεία σε αυτή την έκθεση. Μπορώ να τα συζητήσω λοιπόν απλά αυτά με την εισηγήτρια. Κατά τα άλλα, μ' αρέσει το κείμενο, είναι καλό. Υπάρχουν κάποια σημεία που μοιάζουν τεχνικά, αλλά αν τα κοιτάξετε πιο προσεκτικά θα δείτε ότι υπάρχουν και κοινωνικά, οικονομικά συμφέροντα από πίσω και δεν είναι πάντα εύκολο να βρούμε τη σωστή ισορροπία ανάμεσα στην υγεία, την ασφάλεια, την απασχολησιμότητα και τα οικονομικά συμφέροντα. Αλλά γι' αυτό είμαστε εδώ, για να προσπαθήσουμε να βρούμε την καλύτερη δυνατή ισορροπία. Ο κύριος Στέρκας και μετά ο κύριος Φιλίπ Μπενιόν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μιλώ εκ μέρους της κυρίας Στάινρουκ, που μου άφησε ένα σημείωμα γιατί χρειάστηκε να φύγει και με ενημέρωση και όλες προφορικά για τις τροπολογίες της. Θα ήθελα να σας πω ότι ε, οι σοσιαλιστές γενικά πιστεύουν ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε πως μιλούμε για βασικές προδιαγραφές. Προδιαγραφές και πολύ σημαντικές για την διατήρηση της υγείας των ατόμων που ε, εκτίθενται σε τέτοιου είδους ακτινοβολίες. Δεν είναι πράγματα λοιπόν για τα οποία μπορούμε ελαφρά την καρδία να αποφασίζουμε. Υπάρχουν επιστημονικά, ιατρικά στοιχεία τα οποία ε, είναι ο γνώμονας των αποφάσεων. Το, πρόβλημα δεν το, το βασικό κριτήριο δεν είναι το επάγγελμα, όσο η έκθεση. Γι' αυτό το λόγο πιστεύουμε ότι θα πρέπει να γίνουν μερικέ τροπολογίε έτσι ώστε να προστατεύονται ανεξαρτήτως επαγγέλματο όλοι όσοι εκτίθενται σε ακτινοβολίε πρέπει να λάβουμε άλλωστε υπόψη ότι εμείς δεν πρόκειται να δεχτούμε την οποιαδήποτε μείωση ε, των ορίων χειροτέρευση δηλαδή των υφισταμένων ορίων. Θα πρέπει να βελτιώνεται η προστασία με την νομοθεσία, όχι να ε, υποχωρεί. Δεν είναι σκόπιμο να ε, βρούμε ισορροπίες, να ζητούμε ισορροπίες για οικονομικούς λόγους. Η υγεία ε, ε, είναι ένα αγαθό ανώτερο από την οικονομία. Κατάλληλα συμφωνούμε με την κυρία Μακιντάρ και συμφωνούμε και στα όσα είπε για τους νέους. Υπάρχει και μια ε, τροπολογία σημαντική σύμφωνα με την οποία θα πρέπει να προστατεύσουμε ιδιαίτερα τις εγγύους γυναίκες. Ευχαριστώ. Ε, Κύριος Μπένιν. Ευχαριστώ. Καλωσορίζω την αγνομοδότηση. Η κυρία Μακιντάιρ συνήθως ε, δούλεψε με μεγάλη επιμέλεια. Μην ξεχνάμε ότι είναι μια επικαιροποίηση και ούτω ή άλλως έχουμε ήδη πολύ αποτελεσματικά συστήματα προστασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά κάθε τόσο προφανώς χρειάζονται ε, επικαιροποίηση, ενημέρωση για να λάβουν υπόψη την πιο πρόσφατη επιστημονική γνώση. Και ακριβώς αυτό κάνουμε. Είναι απόλυτα θεμητό και πρέπει να γίνεται κάθε τόσο περιοδικά δηλαδή αυτό το πράγμα. Αλλά αυτό δεν θα πρέπει να μας κάνει να υπερβάλλουμε και να αρχίσουμε να προσθέτουμε διάφορα γραφειοκρατικά θέματα και να φορτώνουμε το κείμενο. Γι' αυτό υπέβαλα κάποιες τροπολογίες για να προσπαθήσουμε να διευκρινίσουμε τις διαφορές ανάμεσα στην, στα συστήματα διοδότησης και καταχώρησης. Αν δεν διευκρινιστεί αυτό, μπορεί να βρεθούμε σε μια περίπτωση όπου θα ζητάμε από τους χρήστες της Ιωνίου ακτινοβολίας να προσπαθήσουν να ζητήσουν εγκρίσεις, άδειες, κάθε φορά που χρησιμοποιούν μια διαδικασία με ακνοβολίες, αντί για μια γενική άδεια, για μια διαδικασία που επαναλαμβάνουν συνέχεια. Προφανώς δεν θέλουμε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Γι' αυτό ακριβώς στην, ε, έχουμε υποβάλει τις τροπολογίες 29 και 30 και ελπίζω να μας το επιτρέψετε με βάση την εντολή μας, γιατί θεωρώ ότι όπως είπε και ο κύριος αυτό επηρεάζει και την ε, ανταγωνιστικότητα και την αποτελεσματικότητα. Πιστεύω λοιπόν ότι οι τροπολογίε αυτέ είναι χρήσιμε. Με ανησυχεί επίση λίγο η τροπολογία 16 που μπορεί να έχει αλυσιδωτές επιπτώσεις ε, αθέλητου χαρακτήρα. Ε, πρέπει να καθίσουμε και να ψάξουμε διάφορα θέματα, γιατί αν δεν προσέξουμε μπορεί να υπάρξουν συνέπειες που δεν ε, θέλαμε να προκαλέσουμε. Το να δημιουργήσουμε, ας πούμε, παραθυράκια από τη μία και γραφειοκρατικά τερατουργήματα από την άλλη είναι αποφεκταίο. Είναι απευκταίο. Ε, θα πρέπει να τα προσέξουμε αυτά τα θέματα. Δεν είναι πολύ μεγάλη σημασία. Και ελπίζω ότι όλοι θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε στο εγγύς μέλλον για αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ. ο κύριος Κλάρκ και στην συνεχεία ο κύριος Κρίστιανσον. Ευχαριστώ. Ο κύριος δίκιο έχει. Αυτό δεν μπορεί να έχει να κάνει μόνο με την απασχόληση. Θα πρέπει να κοιτάξουμε και την πτυχή τη ε, ε, υγείας και τη ασφάλεια. Να είμαστε λογικοί σε ό,τι αφορά τη ρύθμιση Είμαι δάσκαλο και όταν ε, παρουσίασα ιονίζοντα υλικά δεν θα μπορούσαμε να πούμε ότι θα πρέπει να περιορίζεται η ε, χρήση τους, ε, η, η, χρήση τους σε άτομα πάνω των 16. Θεωρώ ότι υπάρχει θέματα σε ό,τι αφορά την έκθεση στην ιονίζουσα ακτινοβολία. Η Διεθνή σε Επιτροπή για την Ιονίζουσα Ακτινοβολία, στην οποία αναφέρθηκε, ορίζει ως ε, γενική σύσταση ένα μίληση ανά έτος για κάθε άτομο. Ωστόσο, κοιτώντα το κείμενο, βλέπουμε ότι στο ε, πρωτότυπο και εδώ πέρα μιλάω για όρια για τους φακούς επαφής, Όχι, το φακούς των ματιών. τους φακούς των ματιών, που προφανώς έχουν μεγαλύτερη ευαισθησία. Το αρχικό κείμενο αναφέρει λοιπόν ότι το επίπεδο θα πρέπει να αποτελεί κατά ανατοτόριο όριο 20 μίλησης το έτος, ενώ η τροπολογία 6 ε, αναφέρεται σε 150, είναι 50, συγγνώμη, ή 15 σε άλλες τροπολογίες αναφέρεται ως όριο. Μίλη Σίβερτς, ανά έτος. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει πιο πολύ έρευνα και να ε, διαβουλευτούμε με τους ε, εμπειρογνώμονες για να βρούμε το σωστό επίπεδο. Σημειώνω ωστόσο ότι το κείμενο αναφέρει και στις αιτιολογίες και σε διάφορα άλλα σχόλια ότι θα πρέπει να γνωρίσουμε ότι το καθεστώς ε, στις διάφορες ευρωπαϊκές ε, χώρες διαφέρει και ότι μία ομοιόμορφη και ε, ομοιογενής προσέγγιση δεν είναι δυνατή και του χρειάζεται ευελιξία σε ό,τι αφορά τους κανόνες και εδώ θα σταματήσω πρόεδρε και κυρία εισηγητρία. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Κρίστενσεν. Ο κύριος Κρίστενσεν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ συνυπέγραψα την τροπολογία για τους frequent flyers, για την κατηγορία των επιβατών που ταξιδεύει πολύ με το αεροπλάνο. Δεν θέλω να δημιουργήσω επιπλέον γραφειοκρατία, αλλά πολλοί κόσμος ε, παίρνει συχνά αεροπλάνο για να δουλέψει για να κάνει τη δουλειά του. Δεν λέω ότι θα πρέπει να δημιουργηθούν και νέοι μηχανισμοί ελέγχου, αλλά όσοι χρησιμοποιούν το αεροπλάνο θα πρέπει να ξέρουν κατά πόσο να ανήκουν σε μια ομάδα υψηλού κινδύνου ή όχι. Αν διευκρινιστεί το θέμα αυτό, θεωρώ ότι θα είναι καλό και φετικό. Ε, Στο η θέλει να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε σας ευχαριστώ για όλα τα σχόλια που λάβαμε και τα μελετήσαμε καλά. Να απαντήσω σε κάποια εξ αυτών. Καταρχάς, ό,τι αφορά την προστασία των ε, επιβατών ε, αεροπλάνων. Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν ε, αυτοί οι frequent flyers, οι οποίοι μπορεί να κάνουν πιο όσες τόσες ώρες όπως και οι πιλότοι στο αεροπλάνο, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να εφαρμοστεί ένα καθεστώς προστασίας, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να εντοπιστεί ένας υπάλληλο ή ένας ε, χώρος εργασίας ο οποίος θα πρέπει να ρυθμιστεί. Για τα πληρώματα είναι πιο απλά τα πράγματα, γιατί ξεκινάμε από τις αεροπορικές εταιρείε και ζητάμε να προστατεύουν το πλήρωμά τους, το προσωπικό τους. Θεωρώ ότι το θέμα αυτό ε, είναι ένα θέμα και πρόβλημα εφαρμογής, σε ποιον θα ζητήσουμε και πού θα ζητήσουμε να εφαρμοστούν αυτέ οι ρυθμίσει. σε ό,τι αφορά τώρα τους ε, μαθητευόμενους και τους φοιτητέ. Αν κοιτάξετε το κείμενο, θεωρώ ότι προβλέπεται προστασία για τους ασκούμενους και σπουδαστές που εκτίθενται σε ιονίζους εκνευολίες κατά την ε, εκπαίδευσή τους, την κατάρτισή τους για τα 16 έτη όριο. Νομίζω ότι η οδηγία είναι σαφής ε, ότι και τα άτομα κάτω τον 16 θα πρέπει να θεωρούνται άτομα του κοινού και θα πρέπει να προστατεύονται ως τέτοια. Τα όρια τώρα για την έκθεση πολλές φορές ε, έχουν αναφερθεί. Η ACRP έχει ε, ζητήσει αυτό το όριο του 1 μιλισίβιτ αναέτος για, τα, για το κοινό. Αυτό αποτυπώνεται και στην οδηγία τα όρια αυτά είναι πιο υψηλά, είναι 30 μιλισιεβίτα ένα έτος για όσους ε, επαγγελματικά έχουν τέτοια έκθεση. Και εδώ και κάποια χρόνια έχουμε 30 αποδεκτικά στοιχεία που καταδεικνύουν ότι ο φακός του ματιού είναι πολύ πιο ευάλωτος, ευαίσθητος από ό,τι θεωρούσαμε. Άρα η Διεθνής Επιτροπή για την Αντιολογική Προστασία προτείνει να περιοριστούν τα όρια τα οποία είχαν ε, προτείνει παλιά από 150 σε 20 μιλισιβίτ ανά έτος. Αυτό και το ακολουθήσαμε ως σύσταση. Τελευταίο θέμα, το θέμα της ε, ομοιομορφίας. Το άρθρο 30 της συνθήκης μας ζητά να δημιουργήσουμε ε, ομοιόμορφα πρότυπα ασφαλείας. Οι υπόλοιπε προδιαγραφέ είναι προδιαγραφέ ελάχιστε. Ευχαριστώ. Η συγκέντρια τηλεγραφικά. Thank you. First of all... Καταρχήν να καθησυχάσω τον κύριο και τον κύριο Θέρκας ότι τα πρότυπα υγείας ε, των εργαζομένων αποτελούν τμήμα των αρμοδιοτήτων μας. Αυτό που προσπαθούσα να διακρίνω είναι ε, το έργο της Επιτροπής Περιβάλλοντος ε, που θα δουλέψει πιο πολύ για το κοινό, το ευρύ και το έργο το δικό μας που εργαζόμαστε πιο πολύ για τα συμφέροντα των εργαζομένων, για την προστασία των εργαζομένων. Έτσι, αυτή είναι η διάκριση που έκανα. Καλωσορίζω την τροπολογία του κ. Μπένιαν. Θα τις υποστηρίξω Η τροπολογία 16 πρέπει να αναθεωρηθεί. Να καθισιάσω τον κύριο Κλάρκ ότι η τροπολογία την οποία μιλάει, η 6, είναι αυτή την οποία απέσυρα. Ε, χρησιμοποίησα την αρχή τα όρια της ICRP που ήταν τα 150 μιλισίβερτ, αλλά αυτά, ε, αυτό το όριο έχει μειωθεί ε, με βάση επιστημονικά δεδομένα, πιο καινούρια, συνεπώς το μείωσα στο 20 το έγγραφό μας επίσης μιλάμε για 16χρονους ως 18χρονους αλλά όχι για πιο νέους. Σας καθησυχάζω και ως προς αυτό κύριε Κλάρκ. Σε ό,τι αφορά τα σχόλια του κύριου Κρίστενσεν για τους τακτικούς επιβάτες θα εξακολουθήσει να είναι ένα θέμα προς συζήτηση. Ευχαριστώ λέει Πρόεδρος. Ωραία θα υιοθετήσουμε την γνωμοδότησή σας αύριο. Το οποίο σημαίνει ότι η Επιτροπή Περιβάλλοντος θα λάβει απόφαση στις 24. Α, στις 20 θα δούμε τους, τις σα σας προτάσεις. Συγγνώμη, έκανα λάθος και στις 21 Μαρτίου θα ψηφίσουμε. Συγγνώμη, λέει η κυρία Περές. Με ανησυχήσατε, δεν Σίγουρα εσείς δεν ανησυχήσατε, αλλά κάποια άλλη μέρη μπορεί να, να ανησύχησαν, να νόμισαν ότι θα ψηφίσουμε αύριο. Επαναρχόμαστε στην, στο σημείο 19 της ημερησίας διάταξης. Λόγω, δίνω το λόγο στον κύριο Κοστέλο. Σχέδιο γνωμοδότησης για τους ε, απόρους. Ε, για τους απόρους. Ο λόγος στην κυρία Κοστέλο. Ευχαριστώ που δίνει το λόγο. Να σας πω ποιο είναι το πλαίσιο αυτής της πρότασης. Να σας, δω, να σας πω τη ποια είναι η φύση του Ταμείου και μετά να ε, κοιτάξουμε λίγο τις τροπολογίες που προτείνω. Σε ό,τι φορά το πλαίσιο. Οι ομιλητές κατά τη διάρκεια της ακρόασης ε, μας είπαν ε, μας μίλησαν για τον αντίκτυπο που έχει κρίση στους πολίτες μας. Και πράγματι χειροτερεύει η φτώχεια και ο κοινωνικό αποκλεισμό σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. 25% του πληθυσμού, 120 εκατομμύρια άτομα δηλαδή, κινδυνεύουν να πέσουν κάτω από το 100% τη φτώχεια. 14 εκατομμύρια είναι πραγματικά άποροι. 10% ζουν σε. Ε, μάλλον 4 εκατομμύρια είναι άστεγοι και πλήττονται κυρίως τα παιδιά. 10% ε, ζουν σε ε, νοικοκυριά χαμηλής εντάσσεως εργασίας. Τα κράτη-μέλη σε περίοδους κρίσης βέβαια δυσκολεύονται να στηρίξουν αυτούς τους ανθρώπους και πράγματι ε, γίνεται πολύ μικρή πρόοδος για την επιτεύξη των στόχων της Ευρώπης 2020. Ε, χρησιμοποιούν το παλιότερα αποθέματα από της παρέμβασης. Ε, ε, τώρα πια συμμετέχουν 20 κράτη-μέλη στο ε, σύστημά μας, το οποίο βασίζεται, όπως σας είπα, σε αποθέματα, γεωργικά αποθέματα. Το σύστημα θα κλείσει φέτος, το οποίο σημαίνει ότι αν δεν αντικατασταθεί θα δημιουργηθεί πρόβλημα στα πιστιστικά προγράμματα σε διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα υποσκαφθεί και η νομιμότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από τη μια μεριά υπαγορεύει λιτότητα και από την άλλη μεριά δεν μπορεί να βοηθήσει τους πιο περιθωριοποιημένους της κοινωνίας μας. Τον Οκτώβριο του 2012 η Επιτροπή πρότεινε ένα σχέδιο κανονισμού για την δημιουργία ενός ταμείου απόρων. Αυτή η πρόταση έχει ευρύτερο πλαίσιο από το προηγούμενο σύστημα ε, θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα των τροφίμων ε, αλλά και γενικότερα θα δώσει βοήθεια σε άστεγους και ε, άπορα παιδιά με μέτρα επίσης κοινωνικής ένταξης. Η στήριξη θα δίδεται στο πλαίσιο εθνικών προγραμμάτων. Τα κράτη-μέλη θα συνεργαστούν με ε, μη κυβερνικές οι οποίες θα εντοπίζουν τους δικαιούχους το Ταμείο θα υποστηρίξει και μια ευρωπαϊκή πλατφόρμα ε, για ε, την αμοιβαία ε, ε διδαχή. Συναντηθήκαμε, με, συναντήθηκα με τους πιο εισηγητές μία φορά και κατηδίαν με κάποιους η Επιτροπή Συνεδρίας και Εξέταση θέμα 23 Ιανουαρίου. Ως αποτέλεσμα έχω 63 τροπολογίες που καλύπτουν μια, ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. Η πρώτη πρόταση που έχω είναι 100% τρόπο ε, χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ η Κομισιόν είχε προτείνει 85% ε, για τα υπόλοιπα κράτη-μέλη, 95% για τα, για τα κράτη που έχουν μνημόνιο. Οπότε εμείς ζητούμε την πλήρη χρηματοδότηση από την ε, Κομισιόν χωρίς η χρηματοδότηση από το κράτος μέλος. Αναφερόμαστε στη σχετική φτώχεια, αναφερόμαστε στην προστασία των δεδομένων και της ιδιωτική ζωής. Θέλουμε να ενισχύσουμε τις συνέργειες, κάτι που είναι πολύ σημαντικό ε, και ελέγχθηκε το Γενάρη στην ακρόαση που κάναμε, συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών, μη κυβερνητικέ οργανώσει κλπ. Ε, επίσης κάνουμε λόγο για συνοδευτικά μέτρα, ε, συνέπεια στο, στους ορισμούς, ενθαρρύνουμε την άρση των εμποδίων στη δωρεά τροφίμων. Για παράδειγμα, μη επιβολή ΦΠΑ, προστασία των, της αξιοπρέπειας των τελικών δικαιούχων και άρση του στίγματος που θα μπορούσε να δημιουργηθεί. Προσπαθούμε να ενισχύσουμε τη σύνδεση με άλλες πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης, δημόσια υγεία ε, και σπατάλη τροφίμων. Επίσης κάνουμε αναφορές στην εκρίζωση της φτώχειας σχετικής με τα τρόφιμα. Σημασία των μελλοντικών δικτύων και αμοιβαία ενημέρωση και μάθησης ε, και υπογραμμίζουμε τη σημασία της αξιολόγησης μέσω έκθεσης που θα υποβληθεί και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχουμε ζητήσει επίσης οι τελικοί δικαιούχοι να είναι δυνατόν να πρέπει να πληρώσουν ένα αντίτιμο, να χρεώνται δηλαδή, αλλά όχι που να μην ξεπερνάει το 10% της εμπορικής αξίας των τροφίμων που λαμβάνουν. Ευχαριστώ πολύ όλους τους και και όλους τους συναδέλφους που έκαναν σχόλια. Ω συμπέρασμα θα ήθελα να πω ότι πρέπει να γνωρίσουμε πως αυτή η πρόταση, αυτό το Ταμείο δεν υποκαθιστά ε, σφαιρικές πολιτικές κατά της φτώχειας. Ε, αυτές αποτελούν ακόμα σημαντική πρόκληση για το μέλλον. Προϋπολογισμός 2,5 εκατομμύρια, λιγότερα από ότι το προηγούμενο πρόγραμμα που είχαμε, ήταν κάτι λιγότερο από 3,1 εκατομμύρια. 2 εκατομμύρια θα είναι δικαιούχοι περίπου ετησίως. 2,5 εκατομμύρια, τα 2,5 εκατομμύρια δεν άλλαξαν από το Σύμβολο Κορυφής ε, που διαπραγματεύθηκε το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Οπότε, παρόλα αυτά όμως, τα 2,5 εκατομμύρια υπολείπονται του ποσού που θα χρειαζόταν για να πετύχει τους στόχους της πρότασης. πρόταση. Παρόλα αυτά η πρόταση ε, είναι θετική και το ίδιο λένε και πολλές από τις μη κυβερνητικές οργανώσεις με τις οποίες ήρθαμε σε επαφή. Ορίζουμε την πρόταση και συμφωνούμε ότι με την πρόταση θα άρουμε κάποια από το, κάποιο από το βάρος της φτώχειας και την, τον αποκλεισμό. Ε, επίσης θα πρέπει να συμπληρώσουμε με, με αυτόν τον τρόπο τις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες. Τέλος, το Ταμείο για τους πιο άπορους είναι μια πρακτική και απτή αναγνώριση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση που θέλει να παίξει το ρόλο της να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της στόχιας και του κοινωνικού αποκλεισμού ε, προσβλέπω στη συζήτηση που θα λάβει χώρα τώρα. Θέλω να ακούσω σχόλια στις τροπολογίες και είμαι στη διάθεσή σας για να τα συζητήσω με τους συναδέλφους. Ε, merci. Chaba, ε, ε, Κύριος Τσάμπα, ο κύριος Όρη και οι υπόλοιποι ομιλητές. Ο κύριος Όρη μάλλον. Ugye ez a jelentés ez azért van előttünk, mert hogy... Τι έκθεση έχει υποβληθεί για αυτή την Επιτροπή. Megszűnik, és ugye rögtön az első probléma itt adódik, hogy a, az... Ε, θέτει ένα πρόβλημα. Η παρέμβαση συνδέεται με άλλα προγράμματα, όπως ας πούμε το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για τα Τρόφιμα, Μιλάμε για 2,5 δισεκατομμύρια, τα οποία ε, μειώθηκαν τώρα στο 1 δις. Ε, αυτά είναι τα νέα που ακούσαμε, αυτά είναι οι φήμες ε, που κυκλοφορούν, αυτές είναι οι φήμες που κυκλοφορούν και ξέρουμε ότι στο μέλλον οι δυνατότητες θα είναι ακόμα πιο περιορισμένες. Συμφωνώ λοιπόν με την εισηγήτρια, την κυρία Κοστέλο, ότι ανεξάρτητα από το πόσο καλά θα εργαστούμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση από αυτού και ως κράτη-μέλη, οτιδήποτε και να κάνουμε, ε, ό,τι και να κάνουμε θα υπολοιπόμεθα σε σχέση με το παρελθόν. Νομίζω ότι είναι προς το συμφέρον μας να έχουμε ένα σύστημα όσο να τον πιο απλό, ε, λιγότερο γραφειοκρατικό, ένα ταμείο το οποίο να μην είναι περίπλοκο, να είναι φιλικό προς το χρήστη, γιατί τελικά ε, υπάρχει ένα έλλειμμα, για να το πω έτσι, και θα το βρούμε μπροστά μας ε, στο μέλλον, παρά τις ε, καλές προθέσεις. Αυτό είναι ξεκάθαρο, έτσι. Τα 2,5 δις λοιπόν ε, υπάρχει πρόβλημα. Καταρχά είναι λιγότερο από ό,τι χρειαζόμαστε, ε, λιγότερο από τι πραγματικέ μα ανάγκε και είναι και ε, λιγότερο από αυτό που έχουν συνηθίσει οι άνθρωποι. για να το πω έτσι. Επίση, δεν ξέρουμε πώ θα επηρεάσει τα επιμέρους κράτη-μέλη και τις κατανομές ε, και τις πιστώσεις ε, για κοινωνικά θέματα που πάνε στους κοινωνικούς τομείς. Ε, και κατά πόσο θα μειωθούν οι συνεισφορές ε, από τους εθνικούς προϋπολογισμούς ε, για τα ίδια θέματα. Αυτή η σχέση δηλαδή του τι δίνουμε εμεί, και τι δίνουν τα κράτη-μέλη θα πρέπει να μας προβληματίσει και εδώ και στο Κοινοβούλιο και στην Κομισιόν και στο Συμβούλιο. Επίσης, η ανάλυση μου συμπίπτει με τη συζητήτρια. Γενικά συμφωνώ με τις προτάσει που έκανε. Νομίζω ότι υπάρχουν σημεία όμως που είναι υπερβολικά λεπτομερή αλλά σίγουρα θα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε με τους σκιώδους εισηγητές όταν συναντηθούμε. Όταν μιλάμε για τη σπατάλη των τροφίμων, για τη σπατάλη των τροφίμων, ναι, πρέπει να καταπολεμηθεί αυτή η σπατάλη. Πρέπει να δούμε τι συνέπειε ε, και να δούμε τι μπορεί να κάνει το πρόγραμμα για να καταπολεμήσει αυτή η σπατάλη. Επίση, ίσω θέλουμε λιγότερη κομισιόν και περισσότερη ε, λειτουργική δράση. Ε, η κομισιόν έχει επαχθεί διαδικασίες για την εποπτεία. Ε, νομίζω ότι καλό είναι να πλουστεύσουμε τι προτάσει που γίνονται για την ε, διαχείριση. Σε ό,τι αφορά την τροπολογία 60, έχω κάποιε αμφιβολίε. Ε, είναι καλή ιδέα αυτό το 10% που ζητάμε από τους άπορους να καταβάλουν. Φυσικά. Αν ζητάς κάτι, υποθέτω ότι κάπως πρέπει να συνεισφέρεις. Από την άλλη όμως, η κατάσταση των ανθρώπων αυτών είναι ήδη κακή, οπότε αυτό το 10% δεν νομίζω ήταν καλή ιδέα. Ε, η Κομισιόν νόμιζε ότι μιλούσε για βοήθεια δωρεάν. Δωρεάν, δωρεάν ήσουν δωρεάν. Α το ξανασυζητήσουμε αυτό το θέμα του 10%. Πάντω, προ το παρόν δεν έχω αποφασίσει, δεν ξέρω αν είναι καλή ιδέα να βάλουμε αυτό το 10% συνεισφορά δηλαδή από του ε, δικαιούχου. Ευχαριστώ την εισηγήτρια ε, για την έκθεση. Θα συνεργαστούμε μαζί της και με τους υπόλοιπους και οδησυγητές. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κάποιες ε, σκέψεις για αυτή την έκθεση και την πρόταση της Κομισιόν. Καταρχάς, χαιρόμαστε που συνεχίζεται μια ευρωπαϊκή δράση για τους ε, πλέον ενδεείς, για τους πιο φτωχούς. Νομίζω ότι βρισκόμαστε σωστό, στη σωστή ατραπό. Μπορούμε να το θεωρήσουμε αυτό, αλλά και με δεδομένο το πολιετές ε, πλαίσιο χαιρόμαστε που, εν πάση περιπτώσει, έχουν γραφεί αυτά τα ποσά, παρότι η συζήτηση για το πολιτές νομικό πλαίσιο δεν έχει τελειώσει. Παρ' όλα αυτά, τα ποσά αυτά έχουν γραφεί ήδη. Ε, δεύτερο, πρέπει να καταγράψω μία απογοήτευση για τα ποσά. Το είπε και η συγγήτρια. Είναι σαφές ότι τα 2,5 δις δεν αρκούν για όλα όσα πρέπει να κάνει αυτό το ταμείο και τη βοήθεια που πρέπει να δώσει στους φτωχούς. Νομίζω ότι πρέπει να συνεχίσουμε τον αγώνα, ούτως ώστε όχι μόνο να κρατήσουμε αυτό το ποσό, αλλά ίσως να προσπαθήσουμε να το αυξήσουμε. Τρίτον, η δουλειά που θα γίνει για τις προτινόμενες τροπολογίες από την εισηγήτρια. Χαίρομαι για κάποιες από τις τροπολογίες. Να τονίσω κάποια στοιχεία. Καταρχάς, η έμφαση που δίδεται ε, στην ε, σχέση με την σπατάλη των τροφίμων ε, φανταστείτε τις το πόσο μπορούμε να υποστηρίξουμε κάποιες τοπικές πρωτοβουλίες, ας πούμε. Ε, εμείς κάνουμε προσπάθεια στην πόλη μου. Είναι σημαντικό θέμα αυτή τη στιγμή της κρίσης, ε, όπου η επισφάλεια για ε, και η ανασφάλεια για όλους αυξάνεται. Επίσης, ε, δίδεται έμφαση στην ανάγκη εταιρικών σχέσεων με τις εθνικές οργανώσεις και τοπικές οργανώσεις. Πολύ σημαντική αυτή η έμφαση. Τέλος, η έννοια της ε, συγχρηματοδότησης. Να την ξαναδούμε ούτω ώστε να μην βάλουμε το τροχοπέδι στη δράση αυτή υπέρ των απόρων. Τελευταίο στοιχείο. Επιτρέψτε μου να καταθέσω και εγώ κάποιες τροπολογίες για να ενισχύσω ακόμα περισσότερο τη σχέση μεταξύ αυτού του Ταμείου, της δράσης και της πρότασης της Κομισιόν και την πλατφόρμα καταπολέμησης της φτώχειας. Φυσικά αυτό το Ταμείο δεν είναι το μόνο μέσο και δεν θα πρέπει να είναι το μόνο μέσο καταπολέμησης της στόχες, αλλά αυτό το μέσο πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι υπάρχει και ένα πλαίσιο ε, στα πλαίσια της στρατηγικής του 2020 και στα πλαίσια αυτά μην ξεχνάμε τον αγώνα καταπολέμησης της στόχες. Μαριάννα Χάρκιν, Καρίν μετά. Κάριν. Ε, υπάρχει κανένα άλλος για να κλείσω τον κατάλογο των ομιλητών. Όχι, Μαριάν Χάρκιν. Ευχαριστώ. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομη. Καταρχά, να ευχαριστήσω την εισηγήτρια γιατί νομίζω ότι έχει κάνει κάποιε εξαιρετικέ ιδέε. Έχει εκφράσει και έχει συμπεριλάβει και τι υποστηρίζω. Τι περισσότερε εξ αυτών δεν πρόκειται να τι κοιτάξω ε, ει βάθο. Τέσσερα σχόλια. Συμφωνώ με το 100% χρηματοδότηση, χωρί η χρηματοδότηση, να ρωτήσω την εισηγήτρια ε, Ποια είναι η άποψή σας για την εθελοντική διαμόρφωση αυτού του, αυτή τη ρύθμιση για τα κρατημέλη, για τα τρόφιμα, για τους άπορους, μιλάμε για μειωμένη χρηματοδότηση. Θα πάνε τα χρήματα αυτά στους πιο ενδεεί. Πείτε μας, αν έχετε ιδέες από αυτού. Μία άλλη ερώτηση ξέρει η συγγήτρια αν υπάρχει μια ενότητα που μπλοκάρει το θέμα αυτό στο Συμβούλιο και μπορεί να κάνει τίποτα η Επιτροπή μας για να ξεμπλοκάρουμε την κατάσταση. Και τέλος. Και πάλι επαναλαμβάνω ότι πρέπει να κοιτάξω την έκθεση καλύτερα, αλλά κάτι που θα κοιτάξω είναι να υπάρχει το απόλυτο ελάχιστο γραφειοκρατίας σας ευχαριστώ πάντως για μια έκθεση καλά ισορροπημένη που περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία. Ευχαριστώ. Κύριε Μαντελή και κυρία Μοργκάντη μετά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ την εισηγήτρια για την προσπάθειά της. Εκ πρώτη όψεως, πέρα από την εμβέλεια αυτού του κειμένου, θα ήθελα να υπενθυμίσω εξ ονόματι της ομάδας μου την στεναρή μας θέση για το σχέδιο προϋπολογισμού για την επόμενη περίοδο προγραμματισμού, όπως προτείνεται αυτή τη στιγμή από το Συμβούλιο. Ακόμα και αν υπάρξει μια προσάυξη τελευταία στιγμή και δοθεί αυτή στο Ταμείο για τους απόρους, το ποσό αυτό είναι ανεπαρκές, αν το συγκρίνουμε, με το τρέχον πρόγραμμα. Και αν, λάβουμε υπόψη την τις νέες προτεραιότητες και τον προεπλασιασμό των προτεραιοτήτων του νέου ταμείου με τα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ δεν θα τα βγάλουμε πέρα. Γιατί δεν λαμβάνονται υπόψη καταρχάς ο προεπλασιασμός της στόχιας και των άστεγων. Αυτό είναι το πρώτο. Δεύτερον, νομίζω ότι είναι και καινή ώρα και κάπου θα πρέπει να υπάρχει σε αυτή την έκθεση μια διάσταση που μας αρέσει εμάς των οικολόγων ε, η πρόθεση των μανάβικων ε, αλληλεγγύης, η αξιοποίηση των τοπικών ε, και ποιοτικών προϊόντων. Με αυτόν τον τρόπο θα, θα, θα καταπολεμήσουμε πιο αποτελεσματικά τη σπατάλη των τροφίπων, θα στηρίξουμε τους τοπικούς γεωργούς, θα αξιοποιήσουμε τις εποχιακές καλλιέργειες και προϊόντα και θα καταπολεμήσουμε την κλιματική αλλαγή λόγω της μεταφοράς των προϊόντων. Γιατί πρέπει να το πούμε και στην Επιτροπή μας στην σε τελική ανάλυση. Και οι πιο φτωχοί έχουν δικαίωμα σε άμεση πρόσβαση σε μια ε, υγιή διατροφή φρέσκια, ε, εποχιακή και ποιοτική. Τέλος. Σε αυτή την έκθεση θα ήθελα να είμαι σίγουρη ότι όλοι οι εταίροι θα εμπλακούν ε, στο πρόγραμμα οι τοπικοί γεωργοί, ε, οι συνεταιρισμοί, ε, οργανώσεις όπως η, τα αλληλέγγυα μανάβικα, ε, οργανώσεις που βοηθάνε τους άστεγους κτλ. Επίσης θα πρέπει να δείξουμε σε ποιο βαθμό η απλούστευση είναι σημαντικό διακύβευμα. Εγώ δεν είμαι υπέρ της χρηματοδότησης. Αυτή τη στιγμή οι οργανώσεις λαμβάνουν άμεσα αυτές τις ε, βοήθειες. Αν ε, βάλουμε τη συγχρηματοδότηση ως προ... προϋπόθεση θα πούν «Α, θέλετε εθνική συγχρηματοδότηση και άρα θα περάσει αυτό το θέμα σε δεύτερη μοίρα, δεν θα είναι προτεραιότητα. Επομένως, θα πρέπει να ξαναδούμε την ιστορία της συγχρηματοδότησης. Και συμφωνώ με τον κύριο Νταρντέν ε, ότι δεν θα καταπολεμήσουμε την φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό μόνο με αυτό το ταμείο. Νομίζω ότι Έφτασε η ώρα και η Κομισιόν και το Συμβούλιο να αναλάβουν τις ευθύνες τους, όπως κάναμε και εμείς εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και να, για να υπάρχει μια πραγματική ευρωπαϊκή στρατηγική για τους άστεγους και για να δημιουργηθεί η Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Καταπολέμησης της Πτώχειας, γιατί όλα τα κράτη δεσμεύτηκαν να μειώσουν τον αριθμό των ενδεών τουλάχιστον κατά 20 εκατομμύρια μέχρι το 2020. Επιτέλους πρέπει να δράσουν, γιατί η φτώχεια και ο αποκλεισμό έχουν ήδη δράσει και έχουν δημιουργήσει ε, ολοένα και μεγαλύτερους αριθμούς ανέργων, φτωχών και άστεγων. Κυρία Μωρά Σαρτιέ, θα επεκτείνω τα όσα είπε η Καρήμα. Είναι σημαντικό να δράσουμε όμως όχι απαραίτητα προς την κατεύθυνση προς την οποία πηγαίνουμε. Χαίρομαι που η συγγήτρια ε, προετοίμασε μια πολύ πλήρη έκθεση. Δεν ήταν εύκολο. Πρώτον διότι μας λείπουν ε, στατιστικά στοιχεία. Η έκθεσή μας ε, υποχρεώθηκε να βασιστεί στα στατιστικά στοιχεία του 2010. Το πρώτο πρέπει να ζητήσουμε σήμερα λοιπόν είναι αυτό. Για μια πραγματική αποτελεσματική πολιτική, προκειμένου να πετύχουμε τους στόχους που έθεσε η Καρύμα μέχρι το 2020, ας υποχρεώσουμε τα κράτη-μέλη να ε, κρα, μα, συλλέγουν στατιστικά στοιχεία. Θα ήθελα λοιπόν να έχουμε στη διάθεσή μας στατιστικά στοιχεία πιο γρήγορα, ε, κατανεμένα αναφύλλω που θα λαμβάνουν υπόψη επίσης την ηλικιακή πυραμίδα των ε, δικαιούχων ε, εμπιστηστικής βοήθειας. Γιατί μιλούμε για αλληλέγγυα μανάβικα, αλλά αυτά βρίσκονται στο πανεπιστήμιο σήμερα. Όλο και πιο νέοι δηλαδή χρειάζονται τέτοιου είδους εμπιστηστική βοήθεια. Πρέπει λοιπόν, πέραν αυτών, πέραν των τροπολογιών που ε, υποβάλει η συγγητρία και της έκθεσης θα πρέπει να ζητήσουμε στατιστικές επικαιροποιημένες που θα μας επιτρέπουν να προσδιορίσουμε τις επιπτώσεις πάνω στις γυναίκες και τις επιπτώσεις πάνω στους, ε, στις διάφορες ηλικιακέ ε, ομάδες. Δεύτερον, συμφωνώ με τα όσα είπε η Μαριάν Χάρκιν για την απαραίτητη ευελιξία. 2,5 ε, δισεκατομμύρια για 28 κράτη-μέλη αυτή τη στιγμή. Ε, αλλάξαμε τρεις φορές την περίμετρο, τη γεωγραφική περίμετρο, η γεωγραφική κάλυψη δηλαδή. Παλότερα ήταν ε, ε, θελοντικής φύσεως. Δεύτερον, ο αριθμός των δικαιούχων αυξήθηκε. Έχουμε περισσότερες χώρες, περισσότερους δικαιούχους και λόγω της ε, κρίσης. Και τρίτον, ε, διευρύναμε και τον τύπο των ε, παρεμβάσεων. Γιατί δεν μιλούμε πλέον μόνο για τρόφιμα, αλλά και για στέγη και συμπεριλαμβάνουμε και την ακραία φτώχεια. Με διανομή ρουχισμού, με ενισχύσεις για πιο ισορροπημένη διατροφή, ε, ενισχύσεις για την υγεία κλπ. κλπ. Συνεπώς αν θέλαμε να πετύχουμε το στόχο μας ε, θα δίναμε στον εαυτό μας και τα άλλα μέσα. 2,5 δισεκατομμύρια δεν είναι αρκετά. Συνεπώς δεν έχουμε το δικαίωμα να γυρίσουμε στο, στα κράτη μας και να πούμε ότι σώσαμε το ταμείο για τους πιο άπορους. Είναι ανεπαρκές αυτό το ταμείο. Το χειρότερο όμως είναι το εξής, ότι το ταμείο αυτό, μάλλον οι πόροι ταμείου από πού προέρχονται, από τους φτωχούς. Γιατί, γιατί χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο εμείς ζητήσαμε το 20% των πόρων του να διατηρηθεί ε, για τα κράτη-μέλη, για την καταπολέμηση της φτώχειας και ο καλύτερος μοχλός καταπολέμησης της φτώχειας είναι η επαγγελματική ένταξη των φτωχών, πρώτος στόχος του Ευρωπαϊκού Ταμείου, και τι κάνουμε, καταστρέφουμε όλους αυτούς τους πολιτικούς στόχους, για τους οποίους είχαμε συμφωνήσει όλοι, και στους στόχους της Ευρώπης 2020 και εδώ στην Επιτροπή, και τώρα τι κάνουμε, τα καταστρέφουμε μέσω των ενισχύσεων, ανεπαρκών ενισχύσεων στους πιο άπορους, πολύ ανεπαρκών ενισχύσεων, δεδομένης της διεύνησης που ε, κάναμε, και τι κάνουμε, παίρνουμε τα χρήματα από τους φτωχού τελικά. Δεν μου αρέσει αυτό. Ξέρω ότι οι φιλανθρωπικές ε, οργανώσεις ε, χαίρονται από την άλλη μεριά ζητούν να κάνουμε περισσότερα, γιατί ε, οι πολίτες ζητούν περισσότερα από τις ίδιες. Ε, εμένα με ενδιαφέρει ιδιαίτερα η συνεργασία μεταξύ των κρατικών αρχών και των τοπικών μη κυβερνητικών οργανώσεων που παρακολουθούν πιο κοντά, από πιο κοντά την κατάσταση. Πρέπει να φροντίσουμε να μην δημιουργηθεί κάποιο μονοπόλιο όλοι να μπορούν να κινητοποιηθούν με συγκεκριμένους πολιτικούς στόχους. Αυτά είναι, αυτές είναι οι δικές μου παρατηρήσεις. Ευχαριστώ την κυρία Κοστέλο για την έκθεσή της. Πολύ καλή η έκθεση, πολύ καλή βάση συζήτησης. Να της πω ότι ανεξάρτητα της πρωτοβουλίας της Κομισιόν, που πρότεινε το κείμενο και ανεξαρτήτως των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που δίνουν την εντύπωση ότι σώθηκαν τα κονδύλια αυτοί που ήταν στο Βερολίνο την Πέμπτη μαζί μου και την Παρασκευή θα αντιλήψαν ότι το θέμα δεν έχει κλείσει, τίποτα δεν είναι σίγουρο. Θα πρέπει να παραμείνουν σε εγρήγορση γιατί η ισορροπία είναι πολύ ανασφαλής, ασταθής μάλλον. Υπάρχει περίπτωση να δημιουργηθεί μια μειοψηφία η οποία θα μπλοκάρει το κοινό συμβούλιο και δεν θα περάσει. Οπότε οι τροπολογίες μας θα πρέπει να συνταχθούν με προσοχή. Δεν θα πρέπει να αλλάξουμε το χρονοδιάγραμμά μας και θα πρέπει να προχωρήσουμε πολύ πολύ γρήγορα. Τώρα θα δούμε πώ στο πολιτευσιο δημοσιονομικό πλαίσιο θα μπορούσαμε να αυξήσουμε λίγο ε, τη χρηματοδότηση του Ταμείου. Ζήτησα από τους συνεργάτες μας να εξετάσουν πού θα μπορούσαμε, από πού θα μπορούσαμε να εξασφαλίσουμε λίγο μεγαλύτερες πιστώσεις. Αλλά ο καθένας από εμά θα πρέπει να πιέσει και τη δική του πολιτική ομάδα. Σε ό,τι αφορά το κείμενο Κοστέλο, ε, έχω και εγώ κάποιες τροπολογίες να προτείνω. Ας προσπαθήσουμε να ε, μην νοθεύσουμε την προσέγγιση μας, τη στάση μας, τη θέση μας. Ε, δικαιούχοι, για παράδειγμα, να δούμε το κατά πόσο θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε ορισμένε ομάδες όπως οι άστεγοι ή τα παιδιά. Ε, για παράδειγμα, ε, πριν, δώσουν τροφή οι δημικές οργανώσεις σε κάποιον ο οποίος είναι προφανώ, φτωχό, θα πρέπει να του ζητούν ε, δικαιολογητικά αποδείξεις. Δεύτερον, Όσοι έχουν δουλέψει με τέσσερα ουρανούς το ξέρουν, ε, αυτές ε, οι, αυτοί οι οποίοι ζητούν επιστημική βοήθεια δεν είναι μόνο αστεγοί και παιδιά. Υπάρχουν ακόμα και φτωχοί εργαζόμενοι και οι οικογένειές τους. Ας μην περιορίσουμε λοιπόν υπερβολικά το πεδίο. Δεύτερη παρατήρηση για το θέμα της συγχρηματοδότησης. Ε, θεωρητικά συμφωνώ μαζί σας. Όμως η συγχρηματοδότηση δεν θα πρέπει να καταστεί υποχρεωτική, αλλά δεν θα πρέπει να απαγορευτεί κιόλα. Ε, ας βρούμε την κατάλληλη διατύπωση που θα μας επιτρέψει να περάσουμε το φίλτρο του Συμβουλίου, διότι με το, με το κονδύλι που προτείνεται δεν θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε τις παλιότερες δράσεις μας. Ο υπεύθυνο στην, ο αρμόδιος υπουργός στην Γαλλία είπε ότι το οποιοδήποτε ευρώ λείπει από αυτό το πρόγραμμα θα το δώσει η κυβέρνηση. Ε, δεν θέλω να τον ε, εκθέσω, ας μην το ξεχνάμε όμως. Η Κομισιόν επίση θα μπορούσε να μας βοηθήσει πώ όλα αυτά θα τεθούν σε εφαρμογή. Να δούμε πώ όλα αυτά θα τεθούν σε εφαρμογή. Γιατί το τρέχον πρόγραμμα κλείνει στις 31 Δεκεμβρίου 2013 και δεδομένων των καθυστέρησεων διαδικασιών θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει το έτος 2014. Υπάρχει περίπτωση να δημιουργηθεί κενό ενός έτους. Θα δώσω το λόγο στην Επιτροπή. Παρακαλώ πολύ, πολύ σύντομα γιατί έχω άλλο ένα θέμα πριν φτάσει ο Επίτροπος. Thank you, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σημείωσα όλες τις προτάσεις και όλες τις συστάσεις. Έχω δει τις τροπολογίες που έχουν κρατεθεί. Προσβλέπουμε και στις καινούργιες. Θα ήθελα τρία σημεία να τονίσω. Καταρχάς, σε ό,τι αφορά την ε, ευελιξία που προτείνει η πρόταση της Επιτροπής ε, και για τον ορισμό της ε, ομάδας στόχου και για το είδος της ε, βοήθειας και της αρρωγής που πρέπει να παρέχεται. Η αρχή της εταιρικής σχέσης είναι μια βασική αρχή για μας και συμφωνούμε απόλυτα ότι οι μη κυβερνητικές οργανώσεις θα είναι οι αντίστοιχες οργανώσεις που θα εφαρμόζουν το μέτρο αυτό. Η ιδέα είναι να ενισχυθούν εφιστάμενα προγράμματα στις χώρες. Όταν είπα ότι η συγχρηματοδότηση θα πρέπει να είναι εθελούσια, θα πρέπει να είναι, τονίζω, σε εθνικό επίπεδο υποχρεωτική. Σε, λαμβάνουμε υπόψη βέβαια τις δυσκολίες που έχουν κάποιες χώρες και γι' αυτό λοιπόν ορίζουμε το 10% ως ε, ποσοστό συγχρηματοδότησης, αλλά η υποστήριξη των εμφιστάμενων μέτρων ήδη υπάρχει από τα κράτη-μέλη. Είναι πολύ σαφής αυτή η αρχή της εταιρική σχέσης με τα κράτη-μέλη. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει ανησυχία για το πώς θα ξεκινήσει η εφαρμογή του προγράμματος. Το συμφωνήσαμε αυτό. Είπαμε ότι θα πρέπει να είμαστε το δυνατόν γρηγορότεροι και ελπίζουμε ο κανονισμός να ε, εγκριθεί το συντομότερο δυνατόν. Το 20% κατανομή εντός ε, του Ταμείου του Κοινωνικού για την κοινωνικό αποκλεισμό δεν συνδέεται με το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τους Άφορους. Ε, το Ταμείο αυτό αποτελεί εξεχωριστή γραμμή ε, του προπολογισμού. Δεν επηρεάζει καθόλου το ποσό που προτείναμε για τον κοινωνικό την κοινωνική συμπερίληψη στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου είναι σαφές ότι τα τρόφιμα αποτελούν σημαντική πηγή για τα άτομα που έχουν στέρηση σε τρόφιμα. Προτείνουμε στον κανονισμό να δημιουργηθούν επιπλέον δίκτυα και υποστήριξη από κράτος μέλος σε κράτος μέλος για να δημιουργηθούν μεγαλύτερες δυνατότητες προκειμένου οι οργανώσεις να έχουν πρόσβαση σε τρόφιμα τα οποία ιδάλλως θα απορρίπτονταν και να έχουμε υπόψη ότι θα πρέπει να είναι καλή ποιότητα τα τρόφιμα αυτά για να μην είναι βλαβερά για τον κόσμο που θα τα καταναλώσει. Μου άρεσε ιδιαίτερα μία παρέμβαση που ανέφερε ότι το ταμείο αυτό δεν υποκαθιστά την συνεκτική σφαιρική στρατηγική για την καταπολέμηση της ένδυας. Μάλιστα, λέει η Πρόεδρος, να είστε πάρα πολύ γρήγορη η εισηγήτρια. Το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό, λοιπόν, γι' αυτό σας δίνω το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, πολλά από τα θέματα θα καλυφθούν μέσω των τροπολογιών. Ε, να αναφέρω σε κάποια θέματα. Το, της χρηματοδότησης του 10%. Αυτό θα είναι εθελοντικό. Πολλές από τις οργανώσεις α, για να διώξουν το στίγμα από τους ανθρώπους θα ζητήσουν από τον κόσμο να πληρώσει 10% κατά μέγιστο. Συμφωνώ με πολλά από τα σχόλια που έγιναν, ιδίω για αυτό περί λιγότερη γραφειοκρατία. Και ξέρω ότι κάνει κάθε προσπάθεια η Κομισιόν, ούτω ώστε να υπάρχει εμπλουστευμένη διαδικασία για το Ταμείο αυτό. Συμφωνώ με τα σχόλια ότι δεν έχουμε επαρκεί στατιστικέ και θα πρέπει να έχουμε πλήρε στατιστικέ. Θα πρέπει να έχουμε ισορροπία μια ισορροπία, δηλαδή σωστέ στατιστικέ και λιγότερη γραφειοκρατία. Η υποστήριξη των μη κυβερνητικών οργανώσεων είναι πολύ σημαντική και η εταιρική σχέση πολύ σημαντικό για τη συγχρηματοδότηση. Συμφωνώ με αυτό που είπε η Κομισιόν, αλλά δεν πιστεύω ότι υπάρχει ανάγκη για συγχρηματοδότηση, γιατί αυτό το ταμείο δεν έχει λόγο ε, να επιβάλλει τη συγχρηματοδότηση που σημαίνει και επιπλέον διοικητικό άχθος. Σύμφωνο, επίσης με όλου του ανθρώπου που είπαν ότι ο προϋπολογισμός είναι ανεπαρκής. Έχουμε περισσότερες χώρε που συμμετέχουν τώρα και άρα επεκτείνεται περισσότερο το Ταμείο. Επομένως υπάρχει ένα θέμα. Και επίσης αυτή η θεροντική συμμετοχή ε, χωρών. Φτάνουμε σε αυτό το σημείο. Αυτό το σημείο είναι σημαντικό μάλλον να πούμε ότι τα λεφτά πρέπει να παραμένουν στο ταμείο. Και αν οι χώρες έχουν opt-out, δεν ξέρω τι θα γίνουν με τα χρήματα. Θα φύγουν τα χρήματα. Είναι ένα θέμα που πρέπει να εξετάσουμε. Και υπάρχει ένα επιχείρημα ότι η Κομισιόν ε, λέει ότι τα χρήματα αυτά δεν είναι για τα κράτη-μέλη, αλλά για τον κόσμο. Ε, σε όλα τα κράτη-μέλη που μπορεί να έχουν πρόβλημα φτώχειας. Επίσης, συμφωνώ με αυτό που υπόθηκε για σκεπτή ξεχωριστή γραμμή προπολογισμού που μπορεί να επηρεάσει το 20% για την ε, κοινωνική ένταξη και κοινωνικό αποκλεισμό. Αυτά, Πρόεδρε, αρκούν. Ευχαριστώ και εσάς και την Κομισιόν για την προθυμία της να απαντήσει στις ερωτήσεις και περιμένω τις τροπολογίες. Θα συνεργαστώ με τους συναδέλφους για να ετοιμάσουμε ένα καλό πρόγραμμα. Και επίσης το ξαναλέω, δεν έχουμε τελειώσει αυτή την ιστορία. Θα πρέπει να δουλέψουμε με ταχύτητα και ελπίζω να περάσει αυτό το πρόγραμμα και ελπίζω να τα καταφέρει και η Ιρλανδική Προεδρία. Μέχρι τις 26 Φεβρουαρίου για τις τροπολογίες 12 το μεσημέρι έχουν προθεσμία. 20-21 Μαρτίου τις εξετάσουμε και θα... στις 22 Απριλίου θα τις εξετάσουμε και θα ψηφίσουμε την ίδια μέρα. Το σημείο 20 έχει αναβληθεί και πάμε τώρα στην εξέταση των 41 τροπολογιών για την έκθεση Τσαμπά Σαγκόρ για την εκπαιδευτική και επαγγελματική κινητικότητα των γυναικών στην Ευρώπη. Κύριε Σόγκορ, έχετε το λόγο. Θα μιλήσω ουγγρικά. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τους συναδέλφους για τη βοήθειά τους και για τις 41 τροπολογίες. Είναι πολύ χρήσιμες. Νομίζω ότι θα συμπληρώσουν την έκθεση και νομίζω ότι γενικά συμφωνούμε. Απλώς δεν μπόρεσα να βάλω όλα τα νέα στοιχεία στην έκθεση όπου αντιμετωπίζουμε την φτωχία, ε, τη φτώχεια, το, την κοινωνική περίθαλψη, ε, τις διαφορές μεταξύ των διαφορών κοινωνικών ομάδων, την ε, κινητικότητα, της μη διακρίσεις ανάμεσα στους διάφορους κλάδους, ε, μη διακρίσεις εναντίον των αναπήρων, ε, γυναίκες, κοινωνικά δικαιώματα, συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας, ένταξή τους στην αγορά εργασίας κλπ. κλπ. Και εγώ έχω υποβάλει δύο τροπολογίες για να βελτιώσουμε την ποιότητα της έκθεσης. Ε, δεν νομίζω ότι θα είναι δύσκολο να φτάσουμε σε συμβιβασμούς. Ε, πολλές από τις τροπολογίες ούτως ή άλλως ε, είναι ταυτόσιμες και άρα θα είναι πολύ απλό να φτάσουμε συμβασμούς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την εισηγήτρια, λέει η κυρία Μπλίνκεβιτσιούτε. Προετοίμασε μια πολύ καλή γνωμοδότηση για την κινητικότητα των γυναικών εγώ παρουσίασα 16 τροπολογίες και πιστεύω ότι μπορούμε να φτάσουμε σε μια κοινή θέση. Όταν μιλάμε για την ένταξη των γυναικών στην εκπαίδευση, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουμε την υγεία, τη φτώχεια, Ιδίω όταν μιλάμε για τις ε, μεγαλύτερες γυναίκες, ε, το θέμα της κινητικότητας των γυναικών. Επίσης μην ξεχνάμε ότι δεν έχουμε ξεπεράσει και δεν έχουμε ρυθμίσει το μισθολογικό χάσμα των δύο φύλων για την ίδια απασχόληση, για την ίδια δουλειά. Επίσης, Ανάλογα με την ηλικία τους ε, και ανάλογα με την κοινωνική τους θέση αντιμετωπίζουν διαφορετικές ε, καταστάσεις οι γυναίκες. Ε, έχουν προβλήματα με χαμηλές συντάξεις. Επίσης οι νέες γυναίκες βρίσκονται σε ιδιάζουσα κατάσταση. Υπάρχει ένα ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24 η Μαΐου του 2012 και το ψήφισμα της 16ης Ιανουαρίου του 2013 όπου ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν την εγγύηση για την νεότητα και νομίζω ότι θα πρέπει να ενθαρρύνουμε και την κινητικότητα των νεαρών γυναικών για εκπαιδευτικού λόγους αλλά και επαγγελματικού λόγους, για την καριέρα τους δηλαδή, και να εξασφαλίσουμε ότι η απασχόληση των νέων γυναικών γίνεται σε υψηλά επίπεδα. Με τις τροπολογίες μου επίσης μιλάω για ένα άλλο σημαντικό σημείο που είναι ε, υψηλά προσόντα για τις γυναίκες, ούτως ώστε και να εκπαιδεύονται, αλλά και να εξασφα... τους εξασφαλίζεται διαβίου μάθηση. Σας ευχαριστώ την προσοχή σε κάποιες από τις τροπολογίες μου. Ε, πιστεύω ότι θα συνεργαστώ με την εισηγήτρια και τους σκιώδης, τον εισηγητή συγγνώμη, και τις σκιώδεις εισηγητές, ούτως ώστε να εντάξουμε όλες τις τροπολογίες. Άλλος κανείς? Όχι. Η Κομισιόν ούτε. Κύριε Σόγκορ, θέλετε να απαντήσετε, όχι. Τέλεια. Τι τέλεια δηλαδή, τέλο πάντων. Είμαστε στην ώρα μας. Στις 20 Μαρτίου θα δούμε τις, τις τροπολογίες, σημαστικές τροπολογίες. Στις 21 θα ψηφίσουμε. Τον Απρίλιο θα ψηφίσει η Επιτροπή Δικαιωμάτων Γυναικών. Τελειώσαμε και με αυτό το σημείο της ημερησίας διάταξης. Διακόπτουμε μέχρι να έρθει ο Επίτροπος. Σα ευχαριστώ. Υπότιτλοι Λοιπόν, συνάδελφοι, προτείνω να ξαναξεκινήσουμε. Ο Επίτροπος ε, κατάφερε να μας βρει. Θέλει να μας παρουσιάσει, σήμερα που υιοθετήθηκε, τη δέσμη μέτρων για την κοινωνική επένδυση. Ένα κείμενο το οποίο το αναμέναμε για πολύ καιρό. Εδώ είναι αυτό το κείμενο. Δεν ξέρω αν στη κάθε σελίδα περιέχει και μία λύση. Πάντως ε, είναι έτσι ένα παχύ έγγραφο. Έχετε το λόγο, Επίτροπε. Ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρησή μου. Χαίρομαι που μπορώ να σας ε, παρουσιάσω αυτό το πακέτο για την κοινωνική επένδυση. Ε, ε, πολυσέλιδο το κείμενο. Σας το παρουσιάζω τη μέρα που υιοθετήθηκε από την Κομισιόν. Ε, χαίρομαι που το Κοινοβούλιο υπογραμμίζει την ανάγκη ενίσχυσης της κοινωνικής διάστασης. Αυτό αναφέρεται και στο, ε, στην, έκθεση Τίσεν, στην έκθεση Γιασλοβιέσκα και στις ε, στην έκθεση Λούπε Φοντανιέ. Το, ιδέσμι για την κοινωνική επένδυση ε, λαμβάνει υπόψη πολλά από τα σημεία των θέσεων του Κοινοβουλίου. Συμπληρώνει τον κύκλο, τον οποίο ξεκινήσαμε ένα χρόνο πριν με τη Λευκή Βιβλία της Συντάξης, συνεχίσαμε με το πακέτο απασχόλησης του Απριλίου 2012, μετά με το πακέτο για την νεότητα το Δεκέμβριο 2012 και τώρα, όλα αυτά μάλλον, ε, τα κείμενα εξυπηρετούν ένα τριπλό στόχο. Είναι πρωτοβουλίες οι οποίες ε, είχαμε αναφέρει στο πακέτο στατικής του 2010, ανταποκρίνονται στην ε, βαθιά οικονομική κρίση και προετοιμάζουν μια πιο στενή, ένα πιο στενό συντονισμό πολιτικών στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι κοινωνικές επιπτώσεις της οικονομικής και χρηματοοικονομικής κρίσης είναι πάρα πολύ σοβαρές. Ο πρόεδρος Μπαρόσο ε, στην, ε, στην ομιλία του για τη κατάσταση της Ένωσης το Σεπτέμβρη μίλησε για, μια, για έναν κοινωνικό συναγερμό. Ε, η ανεργία έχει φτάσει σε πολύ ψηλά επίπεδα, 100, η φτώχεια συγγνώμη, έχει φτάσει πολύ ψηλά, 120 εκατομμύρια πολίτες μας βρίσκονται στο κατόφλι της φτώχειας. Πολύ περισσότερο από παλιά είναι άστεγοι. Αυτές οι τάσεις δεν πρόκειται να αντιστραφούν χωρίς να αλλάξουμε πορεία και προσανατολισμό. Το να βρούμε διέξοδο από την χρηματοοικονομική κρίση είναι σημαντικό. Όμως ο εξυγχρονισμός του, ε, το, του κοινωνικού μας κράτους ε, είναι εξίσου σημαντικός και αυτό προσπαθεί να κάνει το σημερινό πακέτο. Οι κοινωνικές πολιτικές των κρατών μελών θα πρέπει να μάθουν από τα, τα καλύτερα κοινωνικά κράτη της Ευρώπης. Ε, χρειάζεται να είναι πιο απλά συστήματα, να έχουν μια προσέγγιση ε, κύκλου ζωής και να προωθούν την ισότητα. Ε, το πακέτο αυτό περιλαμβάνει ε, μια ε, σύσταση για την καταπολέμηση της φτώχειας των παιδιών, της παιδικής φτώχειας. Το είχαμε ήδη ανακοινώσει δύο χρόνια και δύο μήνες πριν η μείωση των ανισοτήτων από νωρίς, ε, επενδύοντας ε, στην ε, εκπαίδευση και την υγεία των παιδιών, θα πρέπει να είναι βασικό στόχος όλων των κυβερνήσεών μας. Επίσης, υιοθετήσαμε μια έκθεση και κατευθύνσαμε για τις στρατηγικές ενεργού, ενεργού ένταξης με παρική στήριξη του εισοδήματο, αλλαγή στην αγορά εργασίας ε, και υπηρεσίες ε, ε, ποιότητος. Το πακέτο επίσης περιλαμβάνει κάποια αναλυτικά έγγραφα, για παράδειγμα για την άστεγους, την μετανάστευση των σημάτων υγείας, μακροχρόνιες υπηρεσίες υγείας κλπ καλούνται τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιήσουν πιο αποτελεσματικά τον κοινωνικό περιπολισμό που έχουν προκειμένου να απαντήσουν στα προβλήματα της κρίσης. Η Κομισιόν θα παρακολουθήσει στενά τις επιδόσεις των κρατών μελών, των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισής τους ως τμήμα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και θα βελτιώσει τα εργαλεία που διαθέτουμε, για παράδειγμα αναπτύσσοντας προπολογισμούς αναφοράς ε, και υπολογίζοντας την, ε, την ελάχιστη ε, στήριξη εισοδήματος που χρειάζεται. Επίση θα πρέπει να δούμε πώ μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα, κοινωνικά, ε, τα, ευρωπαϊκά κονδύλια, κυρίω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Ε, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο θα μπορούσε, για παράδειγμα, να βοηθήσει ε, στην ε, βελτίωση της, τη ποιότητας κατάρτισης, της ιατρικής και κοινωνικής βοήθειας των παιδιών κλπ. Έχουμε προτείνει τουλάχιστον το 20% των πόρων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου σε κάθε χώρα να χρησιμοποιήσουμε για την προώθηση της καταπολέμησης φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Επίσης προτείναμε το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο να ε, χρηματοδοτηθεί κατά 25% από το, ευρώ, από το ταμείο συνοχής, από τα ταμεία συνοχής. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το θυμηθούμε σήμερα, διότι ε, σύντομα θα ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις μεταξύ Συμβουλίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο σε κοινωνικό επίπεδο το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο είναι το βασική πηγή κοινωνικών επενδύσεων ε, και έχει δυνατότητα μόχλευσης ε, και από, άλλους, ε, και από άλλες πηγές. Το να εξασφαλίσουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο έχει επαρκή επαρκή κονδύλια όπως προτάθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και η βελτίωση των, της αποτελεσματικότητας των επενδύσεών του είναι πολύ σημαντική στόχη. Πρόεδρε, τα Η κοινωνική επένδυση είναι σημείο κλειδί για να βγούμε από την κρίση πιο ε, ισχυρή, πιο ανταγωνιστική, με μεγαλύτερη συνοχή. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να μετακινήσουν ε, ε, την προσέγγιση τους προς την επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό και την κοινωνική συνοχή. Με, αυτό τον, με τις επενδύσεις τώρα θα έχουμε μεγαλύτερο ωφέλη στο μέλλον. Δυστυχώς βλέπουμε παραδείγματα κοινωνικών δαπανών που αποδεκατίζονται ε, ε αλλά αυτό ε, είναι ε, μια στενόμυαλη προσέγγιση. Στο, παρόλα αυτά, στο ε, σημερινό περιβάλλον θα πρέπει να γίνουν συζητήσεις ε, για το ε, κοινωνικό μοντέλο και για την κοινωνική διάσταση της Οικονομικής και Ένωσης παρά την κρίση. Περιμένω θα συνεργαστούμε με το Κοινοβούλιο για να διασφαλίσουμε ότι οι αρχές της Ευρώπης, οι ευρωπαϊκές αρχές για μια δίκαιη και συνεκτική κοινωνία θα διατηρηθούν κύριο Στάρκας όχι. Η κυρία Σαρτιέ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, ευχαριστώ, Επίτροπε, για την ανάλυση σας. Για αυτές τις αναγκαίες κοινωνικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και είπατε ότι μας σας ενδιαφέρει πάρα πολύ οι, κοινωνική, οι κοινωνικές επενδύσεις. Τι σύμπτωση και εμάς το ίδιο. Ξέρετε πολύ καλά ότι εδώ σε αυτή την Επιτροπή, πέρα από τις ε, πολιτικές επιλογές μας, ε, ενδιαφερόμαστε τα μάλα και απαιτούμε στο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο το 25% των, ταμείων, των πόρων των Ταμείων Συνοχής να πάνε για κοινωνικές επενδύσεις ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Για μας είναι το πρώτο αίτημα η πρώτη πολιτική επιλογή που κάνουμε για όλα αυτά τα ταμεία συνοχής. Όταν ακούω τα αιτήματα κάποιων, τα πιεστικά μάλιστα αιτήματα κάποιων κρατών μελών που θέλουν κάποιες επενδύσεις ε, του ΦΕΝΤΕΡ να θεωρηθούν ως επενδύσεις του Ταμείου Συνοχής, μας βρίσκουν παντελώς α, αντίθετους ως μόνιμη συγγήτρια του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου δεν θέλω να πάει το 25% του, του Ταμείου Συνοχής στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Και η δική σας θέληση να υποστήριξετε τις κοινωνικές πολιτικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι ε, και θέληση των υπολείπων να γίνει σεβαστή και να και κυρίως από το σύνολο των κρατών μελών. Επίσης, θα πρέπει να έχουμε την ίδια αποφασιστικότητα, ούτως ώστε το 20% του Ευρωπαϊκού Γεωνικού Ταμείου να πάει ε, για τους πλέον ενδεείς, ούτως ώστε να μειωθεί η μιζέρια. Για μας είναι δύο πολιτικοί στόχοι εκ των όνου με συνεχεία, περιγράψατε με μεγάλη ορθότητα ε, τον προτεσιασμό της φτώχειας. Τα 120 εκατομμύρια Ευρωπαίους, 120 στα 500 εκατομμύρια δεν είναι και λίγα, μεγάλο τμήμα του πληθυσμού. 120 εκατομμύρια που είναι κοντά στο όριο αποκλεισμού και φτώχειας. Και είπατε ότι πρέπει να δράσουμε και να βρούμε μια διέξοδο από την κρίση. Αυτό που μας λείπει είναι μια πολύ ακριβής αποτύπωση της κατάστασης. Και αν θέλουμε να απαιτήσουμε από τα κράτη-μέλη πολιτικές προσπάθειες, οικονομικές προσπάθειες για να μειωθεί αυτή η άκρα ένδια, θα πρέπει να τους ζητήσουμε να δημιουργήσουν αυτές, αυτά τα εργαλεία τα πιλωτικά και τα εργαλεία παρακολούθησης είναι αυτοί οι άνθρωποι αυτοί που είναι απόλυτα ενδεείς, που χρειάζονται επιστημιστική βοήθεια ή που κινδυνεύουν να αντιμετωπίσουν την άκρατη ένδυα. Μιλάμε πολύ για αυτούς. Αλλά πόσοι άντρε, πόσοι, ποια είναι η αναλογία ανδρών και ποσοι ποσοι Ποια είναι η, η ηλικιακή πυραμίδα αυτών που εντάσσονται σε αυτήν την κατηγορία αποκλεισμού και φτώχειας. Η εντύπωσή μας είναι ότι πρόκειται για όλο, ένα και μεγαλύτερα, όλο ένα και νεότερα άτομα. Αλλά αυτά είναι απλές διαστήσεις. Θα θέλαμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλλει στα κράτη-μέλη ένα σύστημα πιλωτικό, ούτω ώστε να έχουμε μια σωστή αποτύπωση της κατάστασης της φτώχειας. Να έχουμε σωστά στοιχεία. Επίσης, μιλήσατε για την αναγκαία κινητοποίηση, ούτω ώστε να αντιμετωπίσουμε την ανισότητα ανδρών και γυναικών. Αυτή τη στιγμή ε, ασχολούμαστε στην επίπτωση ε, της κρίσης στην εργασία των γυναικών. Και εδώ βλέπουμε ότι πρέπει να κινητοποιηθούμε για αυτές τις ανισότητες ανδρών γυναικών, ανισότητες στην καριέρα. Είπατε ότι κάνουμε μεγάλη προσπάθεια για να επενδύσουμε για την εκπαίδευση των παιδιών αλλά θα ήθελα να μιλήσετε και για επενδύσεις σε ισοδύναμες σταδιοδρομίες ανδρών και γυναικών. Ισότιμες σταδιοδρομίες ανδρών και γυναικών. Επίσης, οι αποφάσεις που το στο Συμβούλιο για το Ταμείο Βοήθειας των Πλέον Ενδεών. Νομίζω ότι σήμερα δεν κάνουμε αρκετά για αυτό το θέμα. Και νομίζω ότι δεν είναι η μόνη που το σκέφτεται. 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Ενώ αλλάξαμε πολλές φορές και τις δράσεις αυτού του ταμείου, γιατί θα πρέπει να δώσουμε όχι μόνο επιστημιστική βοήθεια από αυτό το ταμείο, αλλά και βοήθεια για την υγεία, για, τα, για το ρουχισμό, για την υγιεινή, για την καταπολέμηση και την, και την αντιμετώπιση των αστέγων. Δηλαδή, ε, έχουμε 28 κράτη-μέλη, έχουμε πολύ περισσότερες αρμοδιότητες για αυτό το ταμείο και ξέρουμε σίγουρα ότι αυτά τα 2,5 δις δεν αρκούν. Επίσης, ε, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο βλέπουμε τι ποσοστό έχει. Πρόεδρος, ακούστε ποιοι θα μιλήσουν. Ε, Bauer, Άλλος κανείς θέλει το λόγο, εκτός από αυτούς που ακούσατε, κύριε Λάμπερτ. Κλείνω εδώ τον κατάλογο των ομιλητών. Euh, Και, δίνω δυόμιση λεφτά στον καθένα. Ο κύριος Στέρκας. Ο κύριος Στέρκας έχει τρία λεφτά γιατί είναι συντονιστής. Είμαι υποχρεωμένη να το κάνω. Οι υπόλοιποι όμως Δυόμιση λεφτά. Κύριε Θέρκας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ είμαι κατά των προνομίων, αλλά τέλος πάντων θα υποφεληθώ. Ευχαριστώ. Το σωστό είναι να σας ευχαριστήσω για αυτή την πρωτοβουλία που τουλάχιστον στην πολιτική μας ατζέντα αντιμετωπίζει το θέμα των επενδύσεων στην κοινωνία μας. Υπάρχει ένα σύνολο, ένα σύμπλεγμα ιδεών πολύ θετικέ, αναγνωρίζεται το κατεπήγον της κατάστασης, πάθεια και υπάρχουν και κάποια θέματα που τα βλέπουμε για πρώτη φορά. Όπως ένας πολύ σημαντικός για την ομάδα μου συμβιβασμός, ότι δεν θα πρέπει να έχουμε απλώς επαρκή κονδύλια όπως λέει το Συμβούλιο, αλλά θα πρέπει να δούμε και τα νούμερα πολύ συγκεκριμένα. 25 ε, και 20% για την κοινωνική ένταξη. Όλα αυτά, όλες αυτές οι καλές ιδέες όμως δεν συνοδεύονται από δράσεις ανάλογο με το κοινωνικό δράμα που ζουν οι πληθυσμοί μας. Πριν από λίγες μέρες έζησα μία εμπειρία σε μία από τις πιο σκληρές συνοικίες ε, του Παρισιού, στα προάστια του Παρισιού. Όταν βλέπει κανείς αυτές τις καταστάσεις, οι οποίες γίνονται όλο και χειρότερες, το πώς ζει ο κόσμος, ε, πιστεύω ότι πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αυξήσει τα κονδύλια και τις προσπάθειες. Νομίζω ότι όταν αντίθετα μειώνει τις προσπάθειες και τα κονδύλια, ε, είναι σαν να προσβάλλει τους ενδιαφερόμενους, τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις, τους αστέγους κτλ. Δεν είμαστε στο ύψος των περιστάσεων ε, αυτών που ζητάνε οι Ευρωπαίοι πολίτες που είναι θύματα της κρίσης. Είναι σημαντικό να συνεχίσουμε την προσπάθεια, ε, κύριε, Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, ε, εν ώψη του Ιουνίου, ούτω ώστε να υπάρξει ένα πραγματικό κοινωνικό πυλώνα. Να δώσουμε δηλαδή την ίδια σημασία στα κοινωνικά θέματα με τα νομισματικά και τα οικονομικά. Να μην είναι μόνο έγγραφα ε, εργασία και ανακοινώσει, κύριε Επίτροπε. Ε, ενώ η Κομισιόν για τα οικονομικά θέματα προτείνει, επιβάλλει και κυρώνει. για όποιους δεν τηρούν τα πρότυπα, ας πούμε, που προτείνει. Δεν μπορούμε να πούμε στην, στους, πολίτες ότι ε, κάνουμε λιγότερα για τα κοινωνικά θέματα από τα νομισματικά ή τα οικονομικά. Θα πρέπει να είμαστε στο ίδιο επίπεδο. Η επόμενη ομιλήτρια. Ευχαριστώ, λέει η κυρία Μπενά Ράμπα του. Ε, συμφωνώ με τις κοινωνικές επενδύσεις, όπως είπαν και οι συνάδελφοι. Είναι πολύ σημαντική. Αυτά τα ιδέα του, 10, του 25% για τα κοινωνικά θέματα για τις κοινωνικές πολιτικές και υποθέσεις. Είναι πολύ σημαντικό. Η στιγμή, η συγκυρία είναι τρομακτική. Ε, βλέπουμε τον προπολογισμό του Συμβουλίου, τον βλέπουν και οι πολίτες που, είναι, ε, που, πηγαίνει, που κινείται προς άλλη κατεύθυνση. Ε, για μας η τα κοινωνικά θέματα δεν είναι απλώς κόστος, είναι σημαντικός τομέας για επενδύσεις. Δεν μπορούμε να βλέπουμε μόνο τα οικονομικά και νομισματικά θέματα για αυτό το ελάχιστο κατόφλι κοινωνικών δικαιωμάτων και κοινωνικής προστασίας. Στον ΟΗΕ ε, η Επιτροπή Μπασλέ ε, μίλησε για μια ιδέα ότι σε παγκόσμιο επίπεδο θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα, ένα ελάχιστο κατόφλι κοινωνικών δικαιωμάτων. Εμείς δεν θα μπορούσαμε να είμαστε στην πρωτοκαθεδρία, στην αιχμή του, δώρα, η αιχμή Γιατί είμαστε σε αυτή τη θέση, γιατί έχουμε και το, την παράδοση και την ιστορία και τα λοιπά και να δημιουργήσουμε αυτό το κατόφλι. Όταν μιλάω για αυτό το κατόφλι εννοώ για κοινωνικά δικαιώματα. Ε, δεν μιλάω για συντονισμό των κοινωνικών δικαιωμάτων. Έχουμε κοινωνικά δικαιώματα, μπορούμε να τα συντονίσουμε. Αλλά μπορούμε να έχουμε ένα στόχο και διαφορετικές πορείες για να φτάσουμε εκεί. Αυτό ο στόχος να φτάσουμε σε αυτό το βάθρο ας πούμε, κοινωνικών δικαιωμάτων είναι πολύ σημαντικό. Ε, τι γνώμη έχετε γι' αυτό, σας αρέσει αυτή η ιδέα. Επίσης, είναι τρομακτικό ότι έχουμε ε, συστήματα για κάποια κοινωνικά ελάχιστα α, πρότυπα α, που είναι κάτω από το κατόφλι φτώχειας. Δεν θα ήταν λογικό μια πρώτη σύσταση να είναι αυτά τα κοινωνικά ελάχιστα κατόφλια, να είναι τουλάχιστον στο κατόφλι τη στόχιας, τουλάχιστον, ούτω ώστε αυτά τα κοινωνικά ελάχιστα πρότυπα να μας οδηγούν σε ένα εισόδημα αξιοπρεπέ. Εν συνεχεία να έχουμε δράσεις και προγράμματα Γιατί αν δεν το κάνουμε αυτό, στην πραγματικότητα οι δράσει και τα προγράμματα θα είναι εμβαλωματικέ λύσει. Θα, έρθουν να μπαλώσουν απλώ τι τρύπε. Στα κενά του συστήματο προστασία. Σα ευχαριστώ πολύ, η κυρία Μπάουερ. Σα ευχαριστούμε για την ευκαιρία αυτή που μα δίνετε να μιλήσουμε. Τρία θέματα θα ήθελα να θίξω, αν μου επιτρέπετε. Καταρχά, να πω ότι καλωσορίζω το γεγονό ότι μιλάτε για εξυγχρονισμό του κράτου πρόνοια και ότι εστιάζεστε ως επίτροπο στο θέμα αυτό. Ρωτώ πώς ακριβώς σκοπεύετε να το πετύχετε αυτό. Γιατί υπάρχει στην παρούσα φάση μία κοινωνική ένταση, αν θέλετε, και αυτή περιστρέφεται γύρω από το θέμα της απασχόλησης. Πώς μπορεί να επιληθεί αυτή η κοινωνική ένταση, γιατί θα πρέπει να διασφαλίσετε ότι θα πρέπει να ρυθμιστούν και τα θέματα κοινωνικών επιδεμάτων. Κατά δεύτερον, σημειώνω ότι ε, αποδυναμώνεται το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Ε, χάνουμε πόρους. Θα υπάρξει δυνατότητα δημιουργίας συνεργειών, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το Ταμείο για τους πλέον ενδεείς. Μιλήσαμε γι' αυτό πριν από λίγο εδώ στην Επιτροπή. Αναφέρομαι σε όλα αυτά γιατί αναρωτιέμαι κατά πόσον όλα αυτά τα ζητήματα θα χρηματοδοτηθούν από διάφορα προγράμματα. Και το τρίτο θέμα που θα ήθελα να θίξω αφορά τα παιδιά. Θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι τα, οι προτεραιότητέ σα. Θα εστιαστείτε σε πολιτικέ για την εκπαίδευση και την οικογένεια. Πώ πρόκειται να προσεγγίσετε το θέμα αυτό, πώ θα καταπολεμήσετε, με ποια μέτρα θα καταπολεμήσετε την ένδυα των παιδιών στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Μπενιό. Και μετά ο κ. Uh, yes, thanks. Σας ευχαριστώ ορίζω την αρχή ενός ε, πακέτου κοινωνικής επένδυσης. Φυσικά η αποδοτικότητα ενός τέτοιου πακέτου θα κρυθεί από τις λεπτομέρειες και όχι από τον τίτλο. Θα πρέπει να εξετάσουμε τον τίτλο παρόλα αυτά και να δούμε, να εστιαστούμε στη λέξη επένδυση. Δεν θα πρέπει να μιλάμε για πρόνοια με οποιοδήποτε άλλο όρο εξέτασα κάποια προγράμματα στο Birmingham για παράδειγμα, μία από τις πιο δύσκολες ε, υποθέσεις και περιπτώσεις πρόκειται για νέους, άστεχους, που ποτέ δεν έχουν εργαστεί στη ζωή τους και έχουν συνηθίσει πλέον και το γεγονός ότι είναι άστεγοι, τους οποίους ε, τοπικές οργανώσεις τους έχουν δώσει στέγη, τους ε, έχουν εντάξει σε εντατικά προγράμματα για να τους εντάξουν σε δύο χρόνια μέσα στο εργασιακό περιβάλλον. Στα δύο χρόνια συνήθως έχουν βρει δουλειά. Είναι στοχευμένο το πρόγραμμα και είναι μια επένδυση προκειμένου να τους καταστήσει οικονομικά ανεξάρτητους. Αν ε, εξακολουθήσουμε να και μείνουμε σε αυτό το στόχο για να καταστήσουμε τα άτομα τα εξαρτημένα ανεξάρτητα, αυτό θεωρώ ότι αποτελεί επένδυση. Και αυτό θα πρέπει να μας απασχολεί, γιατί με τον τρόπο αυτό έτσι θα συμβάλλουμε πραγματικά στην οικονομική ανάκαμψη. Δίνοντας στα άτομα αυτά τις ικανότητες, τις δεξιότητες που χρειάζονται, τα προσόντα που χρειάζονται, την προσέγγιση στην ε, ζωή που χρειάζονται σε ορισμένες περιπτώσεις μέσω τέτοιων προγραμμάτων. Έτσι θα πετύχουμε και την οικονομική ανάκαμψη, να βρεθούμε σε μια θέση τελικά όπου θα αντιμετωπίσουμε στο μέλλον λιγότερα τέτοια προβλήματα και να σπάσουμε έτσι λοιπόν αυτόν τον φαύλο κύκλο. Όταν θα κοιτάξω τις λεπτομέρειες με την ησυχία μου, ελπίζω να μπορέσω να είμαι πιο συγκεκριμένο στις προτάσεις μου. Καλωσορίζω όμως την προσέγγιση και ελπίζω ότι ο Επίτροπος θα λάβει υπόψη τι προτάσεις μου. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ λέει η Πρόεδρος και τώρα ο κύριος Τσαμπαόρη και μετά η Γιν Λάμπερτ Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ Επίτροπε. Για να είμαι απόλυτα ειλικρινή μαζί σα. Προφανώ. δεν έχουμε εξετάσει ακόμα ολόκληρο το πακέτο, γιατί το λάβαμε σήμερα, αλλά από αυτά που ακούσαμε ως τώρα από αυτά που μας είπε ο Επίτροπος. Η συνολική μου εντύπωση είναι ότι δεν περιλαμβάνονται πολλά νέα στοιχεία στο πακέτο αυτό, ωστόσο θεωρώ ότι είναι ε, στοιχεία τα οποία θα μας βοηθήσουν. Θα βοηθήσουν τα κρατημέλη, θα βοηθήσουν τα, τις υπηρεσίες και θα μας δώσουν και τροφή για σκέψη, αν θέλετε, προκειμένου να αναπτύξουμε ιδέες για τα πιο ευαίσθητα ζητήματα, τα οποία θα πρέπει όλοι να σκεφτούμε. Για να είμαι πολύ ειλικρινής μαζί σας, Ακούγοντα τα εισαγωγικά στα σχόλια, Επίτροπε, μου έκανε εντύπωση το γεγονό ότι μίλησατε για την ε, εξυγχρονισμό του κράτου πρόνοια. Αυτό δεν είναι κάτι το απλό και το σαφέ. Το ξέρουμε αυτό όλοι. Θέλουμε όλοι φυσικά να προστατεύσουμε το κράτο πρόνοια, το ευρωπαϊκό μοντέλο κοινωνικής προστασίας. Δημιουργήθηκε σε άλλες εποχές το κοινωνικό ευρωπαϊκό μοντέλο. Σε άλλες εποχές που ίσχυαν άλλες αναλογίες. Είναι αρκετά λοιπόν ε, επικίνδυνη η κατάσταση, ναι, να εξυγχρονίσουμε το κράτος πρόνοιας, αλλά πώς. Να το σκεφτούμε αυτό από μαζί, τι θα πρέπει να διασωθεί, ποια εργαλεία θα πρέπει να αναπτύξουμε και πού είναι τα αποθέματά μας, τα οποία θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε στο μέλλον. Έχουμε λοιπόν μία βάση ε, Χαίρομαι που αναφέρατε, Επίτροπε, και την παιδική ενδία, Χαίρομαι που μιλήσατε για την διαβίου κατάρτιση και θα επανέλθω σε αυτό. Το καλωσορίζω ιδιαίτερα. Μιλήσατε και για την απασχολησιμότητα. Διάφορα μέτρα προτείνονται προς την κατεύθυνση αυτή. Όλα είναι θετικές προτάσεις. Αν απευθύνεται μια έκκληση λοιπόν προς εμάς να σκεφτούμε όλοι μαζί για το πώς μπορούμε να μεταρρυθμίσουμε το κάτω πρόνοιας, εγώ σίγουρα θα συμμετάσχω και νομίζω ότι όλοι είμαστε διευθυμένοι να το κάνουμε αυτό. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Λάμπερτς. Ευχαριστώ, Επίτροπε. Μία ερώτηση να κάνω. Για θέματα παιδικής ένδυας. Χαίρομαι που το αναφέρατε. Είναι το τελευταίο που αναφέρατε. Μας είπατε ότι το προτιμάζετε εδώ και καιρό. Μιλάτε για την κινητοποίηση των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων. Γνωρίζουμε ότι κάποια κονδύλια ευρωπαϊκά, όχι ίσως της Επιτροπής μας, αλλά κάποια κονδύλια έχουν ως στόχο, στο τους, ένταξη των ε, Ρωμά και ότι κάποια από τα εργαλεία αυτά δεν έχουν αξιοποιηθεί. Θα ήθελα λοιπόν να μας πείτε πώς η υπηρεσία τη Επιτροπή θα συνεργαστεί με τι άλλε υπηρεσίε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου οι συστάσει αυτέ να έχουν αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά την παιδική φτώχεια σε ό,τι αφορά και την κινητοποίηση των υφιστάμενων κονδυλίων για να πετύχουμε του κοινού μα στόχου, Γιατί ένα από τα θέματα που αναφέρθηκε είναι ότι υπάρχουν διάφορε μορφέ, πολλαπλέ μορφέ ένδυα, πολλαπλέ μορφέ διακριτική μεταχείριση. Πώ λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εσεί θα συνενώσετε, θα συγκεντρώσετε όλες τις δυνάμεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να πετύχουμε τους στόχους που έχουν τεθεί στις συστάσεις. Thank you much, uh, first of all, for the, uh, the, the kind... Uh, Καταρχήν ευχαριστώ πολύ για τη θερμή υποδοχή και για τα καλά σας λόγια. Ευχαριστώ πολύ και για τις ερωτήσεις. Όπως είπε ο κ. Μπένιαν, ο τίτλος είναι σημαντικός. Ο τίτλος, μπορώ να σας πω, ήταν ήδη επιτυχία από, το, από πέρσι το καλοκαίρι, όταν τον πρώτο χρησιμοποίησαμε, όταν ξεκινήσαμε να δουλεύουμε αυτή την πρωτοβουλία στην Κομισιόν. Ο τίτλος ήδη υποδεικνύει την ε, διάθεση ανανέωσης, τη διάθεση να κοιτάξουμε προς το μέλλον την κοινωνική πολιτική. Όταν δείτε τις λεπτομέρειες θα το καταλάβετε. γιατί χρειάζεται αυτή η προσπάθεια εξυγχρονισμού. Ε, είναι πολύ σημαντικό αυτό, είναι πολύ σημαντικό στόχος για τον εξής λόγο. Πώς είπε ο κύριος Όρη, πολλά από τα συστήματα κοινωνικής προστασίας ε, γεννήθηκαν μετά τον πόλεμο, μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο Η εξέλιξη όμως των οικονομικών συστημάτων, Ευρωπαϊκή Ένωση, παγκοσμιοποίηση, τελικά και η οικονομική κρίση ε, δημιούργησε προκλήσεις σε αυτά τα συστήματα. Αυτές οι προκλήσεις είναι και ευκαιρίες βέβαια ταυτόχρονα. το να μιλάμε για παράδειγμα για ε, έναν μακρύτερο κύκλο ζωής, ένα μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής είναι πολύ σημαντικό. Πάντως το κοινωνικό κράτος ορίζεται και προσδιορίζεται σε εθνικό επίπεδο. Πλην όμως σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουμε τη δήλωση δικαιωμάτων μεταξύ αυτών και των κοινωνικών δικαιωμάτων και επίσης ε, διαθέτουμε και κάποια εργαλεία που μπορούν να υποστηρίξουν την καλύτερη λειτουργία των κοινωνικών κρατών. Και ως απάντηση στην κρίση ενισχύσαμε επίσης και την οικονομική διακυβέρνηση που μπορεί να ισορροπηθεί, να εξισορροπηθεί μόνον ε, αν αντιμετωπίσουμε και τις κοινωνικές προκλήσεις ε, προσπαθώντας να βοηθήσουμε τα κρατημέλη να λύσουν τα σχετικά προβλήματα ταυτόχρονα με την επίλυση των οικονομικών και γενικότερα μακροοικονομικών προβλημάτων τους. Οπότε πρέπει να συμπληρώσουμε αυτό το κοινό ανάμεσα στην δήλωση περί δικαιωμάτων και κοινωνικών δικαιωμάτων και της ύπαρξης εργαλείων αφενός και από την άλλη μεριά της αρμοδιότητας των κρατών μερών για την κοινωνική πολιτική. Με τρεις τρόπους μπορούμε να κλείσουμε αυτό το κενό, να το καλύψουμε. Πρώτον, να ενισχύσουμε την ανοιχτή μέθοδο συντονισμού, δηλαδή τη μεθοδολογία κατά βάση της ε, ε, διαδικασίας αυτής. Για παράδειγμα, να βελτιώσουμε το σύστημα των δικτών, το benchmarking, για προκειμένου να κάνουμε σωστές επιλογές στην κοινωνική πολιτική συμπεριλαμβανομένων και των οικονομικών επιλογών μετά την εμπειρία της χρήσης των εργαλείων που έχουμε να την εκμεταλλευτούμε έτσι ώστε να χρησιμοποιηθεί από τις χώρες και από τις περιφέρειες οι οποίες ακόμα δεν κάνουν χρήση. Το έγγραφο επίσης ε, ορίζουμε, μιλούμε για το πώς θέλουμε να εντάξουμε στην οικονομική διακυβέρνηση θέματα όπως η φροντίδα των παιδιών και διάφορα άλλα. Απασχόληση των γυναικών. που ήταν εκεί τα τελευταία δύο χρόνια, αλλά με αυτό το πακέτο έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε συστηματικά με το Κοινοβούλιο, με το Συμβούλιο και με άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, εμπλεκόμενους φορείς, ε, πώς το ευρωπαϊκό εξάμεινο μπορεί να συμπεριλάβει και αυτά τα κοινωνικά θέματα. Εξυγχρονισμός σημαίνει επίσης και διάφορα άλλα στοιχεία. πανεπιστημιακοί εμπειρογνώμονες μας βοήθησαν και πιο συγκεκριμένα τη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης να αναπτύξουμε το πακέτο του πακέτου και το βασικό ζήτημα, το light motif ήταν γιατί οι σκανδιναβικές ε, χώρες έχουν πετύχει ε, σε σχέση με πολύ περισσότερο από τι άλλες και τι μπορούμε να μάθουμε από την εμπειρία τους. δεν δείτε τις λεπτομέρειες του πακέτου, έχουμε προσδερήσει τι είναι αυτό το οποίο μπορεί να αντιγραφεί. Τέτοιου είδους ε, επιχειρήματα, τέτοιου είδους ε, ερωτήματα και απαντήσεις εμφανίζονται σε όλο το κείμενο του πακέτου που υιοθετήσαμε. Απαντώ στην κυρία Μπάουερ να πω το εξής. Ε, Η αιρεσιμότητα είναι κάτι καινούριο. Ορισμένες από τις κοινωνικές ενισχύσεις μπορούν να υπόκεινται σε αιρεσιμότητα. Το, αυτό το είδαμε και στις σκανδιναβικές χώρες, το έχουμε δει. Ε, ας είμαστε ειλικρινεί. Ε, ακόμα και στην Βραζιλία και σε άλλα μέρη του κόσμου, ε, χρησιμοποιώντας την αιρεσιμότητα, έχουν εφαρμοστεί ε, πολύ επιτυχή προγράμματα κατά της φτώχειας. Ε, η αιρεσιμότητα μπορεί να συμπληρώσει, όχι να αντικαταστήσει ε, εργαλεία τα οποία έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δυο λόγια για τα χρηματοοικονομικά μέσα και εργαλεία. Ευχαριστώ την κυρία Μωρέν Σαρτιέ για την υποστήριξή της και τις προσπαθίες της για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Νομίζω ότι η διαφορά είναι, θα είναι τεράστια αν ε, χρησιμοποιήσουμε εργαλεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για παράδειγμα, η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων και η βοήθεια για τους απόρους έχουν οριστεί με τρόπο που θα γίνει προβληματικός αν δεν ε, ξεκαθαρίσουμε τον ορισμό του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Συνεπώς, πρέπει να οριστεί το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Επίπεδο σε ε, επίπεδο ευρωπαϊκή Ένωση. Και με αυτόν τον τρόπο και το Κοινοβούλιο θα μπορεί να το ελέγξει καλύτερα σε σχέση με το αν το Ευρωπαϊκό Ταμείο παραμείνει ως υπόλοιμα, ως ε, υπόλοιματικό ταμείο. Ε, καταλαβαίνω ότι μακρηγορώ, αλλά θα έχουμε και άλλες ευκαιρίες να τα ξανασυζητήσουμε. Ευχαριστώ πολύ για την πρώτη αυτή ε, πολύ επικοδομητική και ουσιαστική συζήτηση. Ευχαριστώ που ήρθατε. Την ημέρα που υιοθετήθηκε το κείμενο. Φυσικά θα έχουμε και άλλες ευκαιρίες να το συζητήσουμε. Είναι μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων σήμερα.